the choices we have presented in our campaign are really Είναι τώρα πολιτικές ε, επιλογές. Το θέμα είναι τι πολιτικό χρώμα θα θέλατε να έχει η Ευρώπη μετά τις εκλογές. Επομένως, το μήνυμα με το οποίο πηγαίνουμε στις εκλογές είναι έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ποιος θα κυβερνήσει την Ευρώπη. Είναι η δική σας ψήφο που θα κάνει τη διαφορά. Είναι οι πρώτε εκλογέ οι οποίε γίνονται μετά από τη συνθήκη τη αγώνα, την εφαρμογή τη, Για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκλέξει τον πρόεδρο τη Κομισιόν, δεν θα τον επικυρώσει, δεν θα τον προτείνει, θα τον εκλέξει. Για πρώτη φορά τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη έχουν ε, παρουσιάσει επικεφαλής ψηφοδελτίων που είναι στην προεκλογική εκστατεία. Έχουμε πέντε λοιπόν επικεφαλής ψηφοδελτίων που αγωνίζονται για να κάνουν ορατές τις προεκλογικές εκστρατείες των κομμάτων τους. Έχουν διοργανωθεί διάφορες συζητήσεις μεταξύ των υποψηφίων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει παίξει ένα πρωτοπόρο ρόλο στην προετοιμασία αυτών των συζητήσεων, των debates. Έχει διοργανώσει και μία συζήτηση μεταξύ των πέντε υποψηφίων που θα είναι η πιο σημαντική. Ίσως γιατί θα είναι η μόνη που θα έχει και τους πέντε υποψηφίους, θα λάβει χώρα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα στις 15 Μαΐου. Και θα είναι μια <clears throat> συζήτηση που θα οργανώσουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση Τηλεοπτικών Καναλιών, την EBU, και θα υπάρξει αυτή η συνεργασία φυσικά και με εθνικά κανάλια, εθνικά τηλεοπτικά κανάλια. Για παράδειγμα, για να σας δείξω το πόσο έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση και έχουμε αφιερώσει πάρα πολλούς πόρους στο να είμαστε πιο κοντά στα μέσα ενημέρωσης, γιατί για μας τα μέσα ενημέρωσης παίζουν ένα προεξάρχοντα ρόλο σε αυτή την προεκλογική εκστατεία πληροφόρησης. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα επίσης γιατί βλέπουμε το πώς τα μέσα ενημέρωσης και ο τύπος έχουν ανταποκριθεί στην εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα. Έχει πολύ πιο πολιτικό χαρακτήρα η συζήτηση. Εστιάζεται περισσότερο στις θέσεις και όχι τόσο πολύ όσο στο παρελθόν, με κάποιες εξαιρέσεις ίσως, στα, δεν εστιάζεται σε σκάνδαλα ή σε ε, σπατάλες χρήματα. Η συζήτηση λοιπόν η οποία έχει αναπτυχθεί είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται όλο και πιο ορατή. Και τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση εκλογέων στις ευρωεκλογές από ό,τι στο παρελθόν, την τελευταία, στις εκλογές του 2009. Δεν είναι αυτός ο μόνος μας στόχος φυσικά, η μεγαλύτερη προσέλευση των εκλογέων, αλλά αν όλα τα, όλοι οι εμπλεκόμενοι, τα πολιτικά κόμματα και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί μπορούν να κινητοποιήσουν την κοινή γνώμη, ίσως θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια καλύτερη Ευρώπη για ένα καλύτερο μέλλον και για καλύτερη δουλειά από κοινού και καλύτερη ζωή για όλους. Είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα έρθει αργότερα θα σας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλύτερα από μένα μπορεί να σας παρουσιάσει το πολιτικό πλαίσιο και το γιατί αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά και γιατί για σας είναι τόσο σημαντικό να κατανοήσετε γιατί η δύναμη που έχει ο τύπο και τα μέσα ενημέρωση εν γέννη μπορούν να χρησιμοποιηθούν εποφελώ στι ευρωεκλογέ. Απλώ θα ήθελα να ε, συμπροεδρεύσω στην σημερινή πρωινή συνεδρίαση μας με τον κύριο Λιπόλ από την Κομισιόν, τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά η διαθεσμική συνεργασία ήταν πραγματικά μια μεγάλη επιτυχία και με τον τρόπο αυτό γίνεται σαφές ότι τα θεσμικά μας όργανα έχουν ε, κατά κάποιο τρόπο ανδρωθεί. Έχουμε κατανοήσει ότι οι ευρωεκλογέ δεν είναι μονάχα ένα ραντεβού που δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε πέντε χρόνια, αλλά είναι ένα κοινό εγχείρημα, είναι μια κοινή προσπάθεια, ένας κοινό στόχος για να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να υπάρξει και καλύτερη συνεργασία, όλα αυτά προς όφελος του πολίτη, γιατί η Κομισιόν, το Συμβούλιο και η Κομισιόν μπορεί να είναι λιγάκι απόμακρα, αλλά για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο έχει με τη συνεργασία των τριών θεσμικών οργάνων συνεργαστεί εδώ στις Βρυξέλλες και στα κράτη-μέλη μέσα από τα γραφεία πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις ε, αντιπροσωπείες της Κομισιόν και από τους ε, εκπροσώπους τύπου της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Γίνεται λοιπόν αυτή η προσπάθεια να υπάρξει μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση και με τη βοήθεια των εθνικών αρχών. Ε, Γκρέγορη λοιπόν με μεγάλη χαρά μπορώ να σου δώσω τον λόγο και ελπίζω ότι δεν θα ε, διαψεύσεις όλα αυτά τα οποία έχω πει ότι συνεργαζόμαστε τόσο καλά μαζί. Όχι, όχι, με τίποτα, με τίποτα, γιατί συνεργαζόμαστε άριστα. Και εγώ όπως και η Χουάνα, σας ευχαριστώ, καλώς ήρθατε στις ε, Βρυξέλλες και ακριβώς το ότι βρίσκεστε εδώ σημαίνει ότι ενδιαφέρει η Ευρώπη. Δεν είναι σημαντικό. Ακριβώς ε, απλό ενθουσιασμός αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το ότι σας νοιάζει θέλετε να έρθετε εδώ στην καρδιά της Ευρώπης και θέλετε εδώ να συζητήσετε, να συζητήσετε με εκείνους οι οποίοι εργάζονται στις Βρυξέλλες. Στι ε, στις όπου πολλές φορές είναι συνώνυμο της Ευρώπης, όπως χρησιμοποιείται για αυτόν τον τρόπο και να ξεκινήσουμε να, ακούσετε από μέσα το τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα έρθει και ο Γενικό Γραμματέας και θα μπορέσετε να υποβάλλετε ερωτήσεις, θα μπορέσετε να προκαλέσετε τις αντιδράσεις αυτών των ανθρώπων που δουλεύουν από τα μέσα. Οπότε ε, δεν θα με γνωρίσω, απλώς θέλω να σταθώ σε τρία σημεία. Πρώτα πρώτα θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα πιο βασικά, στις πιο βασικές αξίες, στις κοινέ αξίες που είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό ούτως ώστε να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία των ε, ΜΜΕ για να υπάρχει πλουραλισμός και οπότε θα πρέπει μαζί να ε, δούμε πώς θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις ε, πηγές ε, που έχουμε πολλές πηγές για τη δουλειά σας και αυτό να αφορά και ρεπορτάζ για την Ευρώπη. Πρώτα πρώτα να σας πω ότι είμαι ο Διευθυντής για τα θέματα επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενικός Διευθυντής αυτής της Γενικής Διεύθυνσης που δεν ενδιαφέρεται μόνο ε, στο να σας παρουσιάσει μια ρόδινη εικόνα. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να ε, εξασφαλίσουμε το ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα ακούσετε τις λεπτομέρειες των θεμάτων και από τους άλλους ομιλητές σε λίγο, γιατί έχει σημασία η Ευρώπη και γιατί αυτή τη φορά όλα είναι διαφορετικά από ό,τι ε, στις προηγούμενες ε, ε, ευρωεκλογέ και γιατί έχει σημασία το τι θα ψηφίσει ο κόσμος αλλά είναι σημαντικό να ασκεί στο το δημοκρατικό του δικαίωμα να μπορεί να λάβει αποφάσεις βάσιμες, λογικές και αυτό είναι ευθύνη δική μας και δική σας. Και έρχομαι τώρα στο πρώτο σημείο που θέλω να αναπτύξω, τον πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης που είναι μια κοινή αξία εδώ στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο της ειρήνης και της δημοκρατίας για περισσότερο από έξι δεκαετίες. Βεβαίως, ε, που και που έχουμε κάποιες κρίσεις που ξεσπάνε, όπως έχουμε αυτή τη στιγμή την ε, κρίση που σοβεί στα ρωτολικά μας σύνορα και βλέπετε ότι εκεί πέρα η έλλειψη ελευθερίας των ΜΜΕ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Άρα πλουραλισμός και ελευθερία των μέσων είναι η καρδιά κάθε δημοκρατίας και εσείς αποτελείτε την απόδειξη. Ρίξτε μια ματιά δεξιά, αριστερά σας και θα δείτε ότι σήμερα το ακροατήριό μας ε, αντιστοιχεί σε αυτό που λέμε σαν σύνδεμα για την Ευρώπη, ενωμένη στην πολυμορφία, ενωμένη στο ότι ενδιαφερόμαστε, νοιαζόμαστε για την Ευρώπη και πολυμορφία, μια που ε, όλοι εδώ προερχόμαστε ο καθένας από άλλη χώρα, έχουμε διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική γλώσσα χρησιμοποιούμε και επίσης εκπροσωπούμε και διαφορετικά μέσα ενημέρωσης, τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα και μόλις το 1950 είχαμε την ε, ε, Σύμβαση Ανθρωπινών Δικαιωμάτων, οπότε και κατοχυρώθηκε αυτή η, ελευθερία του να διατυπώνει κανείς τη γνώμη του, να μπορεί να δώσει ή να λάβει πληροφορίες χωρίς να παρεμβαίνει κάποια δημοσία αρχή και αυτό κάτι να ξεπερνά τα σύνορα σαν ε, αρχή. Και από τότε το έχουμε επαναδιατυπώσει επανειλημμένα σε διάφορα έγγραφα ε, που έχουν ενσωματώσει ε, αυτά τα θεμελιώδης αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό αφορά και σε νόμους που έχουν θεσπιστεί γιατί σύμφωνα με το κοινωτικό δίκαιο θα πρέπει να δίνονται εγγύσεις για αυτά τα σχετικά δικαιώματα. Έτσι σύμφωνα με τους ε, reporter ε, χωρίς σύνορα ισχύουν αυτές οι αρχές στην Ευρώπη όπως βλέπουμε από τα δημοσίευτους και ε, έχουμε τις 50 κορυφαίες χώρες που σέβονται την ελευθερία και σε αυτές τις 50 χώρες συμπεριλαμβάνονται όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να δρανούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πασκαρτίνο των Συνθήκων παρακολουθεί προσεκτικά το αν τα κρατημέλη τηρούν το κοινωτικό δίκαιο το οποίο, είμαστε, το οποίο πρέπει να εφαρμόζουμε. Πάντως το κοινωτικό δίκαιο θα έχει νόημα εάν δεν ασκούσετε εσείς ε, το δικό σας λειτουργήμα και να ασκείται μια δημοσιογραφία υψηλού επίπεδου σε όλη την Ευρώπη. Να ενημερώνει το κόσμο για τα ενδιαφέροντα θέματα, να συνδυάζετε διαφορετικές πηγές, να μπορείτε να ακούσετε διαφορετικές γνώμες, να έχουμε έτσι την συνέργεια και μέσω της οποίας αυτό που δεν μπορεί να κάνει μια χώρα μόνη τη, τα κάνουν οι χώρε από κοινού. Πάμε τώρα στι ε, πηγέ των πληροφοριών. Ξέρω ότι ε, είστε ενήμεροι γι' αυτό, απλώ σα υπενθυμίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορείτε εσείς να έχετε πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες, στην πρώτη ύλη ούτως ώστε να μπορείτε να έχετε τις πηγές που θα σας επιτρέψουν επαγγελματικά να δουλέψετε. Πρόκειται για πληροφορίες από πρώτο χέρι δηλαδή. Πρώτα πρώτα έχουμε την υπηρεσία για τα οπτικοακουστικά που δίνει τις φωτογραφίες. Δεν υπάρχει εκεί editing, οπότε αυτό είναι η πρώτη ύλη για σας να τα χρησιμοποιήσετε και αυτά να φτάσουν στους ε, τηλεθεατές, ακροατές, αναγνώστες. Αν θέλετε κάποια πληροφορία, θέλετε κάτι να ρωτήσετε σχετικά με αυτό, μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες μας. Και εδώ έχουμε την, τον ε, Αλέον Τιμό από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος είναι στη διάθεσή σας, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε για αυτές τις πηγές πληροφοριών που υπάρχουν. Το, το τελευταίο που θέλω να σας ε, αναφέρω είναι το ότι θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να χρησιμοποιήσετε όσο μπορείτε καλύτερα όλες αυτές τις ε, πληροφορίες για την Ευρώπη και με υπευθυνότητα να δίνετε μία εικόνα ε, σφαιρική, ολοκληρωμένη. Και όχι μόνο επειδή τώρα αυτέ οι ευρωπαϊκέ εκλογές είναι διαφορετικέ αλλά και, γιατί και για σήμερα και για το μέλλον η Ευρώπη είναι πάρα πολύ ε, σημαντική τις μέλουσε γενναίες και έχει σημασία και για τις Βρυξέλλε και για όλη την Ευρώπη ε, ας πούμε οι Ουκρανοί σε εμά ε, προσβλέπουν και ε, το, ο πλούτος εδώ που υπάρχει είναι το μισό του ΑΕΠΟΛ του κόσμου. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή την προβληματική που θα πρέπει πάντοτε να βασίζεται σε κάποια ε, δεδομένα, σε, να είναι τεκμηριωμένη. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και εμείς στην Γενική Διεύθυνση για την Επικοινωνία. Συμβουλεύουμε, μιλούμε, αλλά κυρίως ακούμε. Και αυτό και θα κάνουμε σήμερα εδώ περιμένουμε πώς και πώς να σας ε, ακούσουμε. Ε, η Ευρώπη πάντοτε πρωταγωνιστής στις ε, ειδήσει, άλλες φορές είναι από διοπομπέως τράγος, αυτό κάνουν οι κυβερνήσεις, όταν κάτι πάει στραβά κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατηγορούν τις Βρυξέλλες. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ίσως αυτή η τάση θα έπρεπε να αντιστραφεί και προς τούτο χρειάζεται ο κόσμος να είναι ενήμερο για τα επιτεύγματα πάντως. Ο ρόλο των μιμήσεων είναι το να έχουν κριτική στάση. Οπότε γι' αυτό λοιπόν, πρέπει να χαιρετήσουμε αυτό σα το ρόλο. Και σήμερα επομένω θα πρέπει να συζητήσουμε και να δούμε ποια είναι η αλήθεια για το τι γίνεται στι Βρυξέλλες, πώ έχουν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε σα εύχομαι να έχετε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστώ. Αν δεν σας πειράζει θα ήθελα να ζητήσω από τους δημοσιογράφους να κάνουν τις πρώτες ερωτήσεις ενώ περιμένουμε τον κύριο Κλάσουελε. Τόργετέλα, λέγομαι συντάκτη στην ε, Δανέζικη τηλεόραση, καλύπτω από το 77 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως ξέρετε, στην Ευρώπη υπάρχει έντονος σκεπτικισμός, τουλάχιστον στη χώρα μου. Ένα από τα ερωτήματα στη χώρα μου είναι ο προϋπολογισμός και ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε πάνω από 100 δημοσιογράφοι εδώ. Βλέπω 7 ε, να χρησιμοποιούν ακουστικά. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι γιατί χρειάζεται η διερμηνία. Όπως είπα καλύπτω το Κοινοβούλιο το 1977, γνωρίζω πως ε, όλοι οι άνθρωποι εκεί πίσω από το γυαλί είναι πολύ ικανοί, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αλλά μια που έχουμε κρίση στις ε, ευρωπαϊκές ε, χώρες, ε, οι οποίες κάνουν οικονομία όπως και οι εταιρείε. Εδώ όμω προφανώς χρησιμοποιείται λεφτά σε πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι θα μας πείτε, τι μπορούμε να πούμε στους θεατές μας, τους συνδρομητές μας για το τι, μπορείτε, τι κάνετε για να κάνετε οικονομίες στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. I'm sorry because um, I think that Ο ήχος, ο ήχος ε, δεν λειτουργήσε. Αλλά νομίζω την ερώτηση μπορεί να την απαντήσει και ο φίλος μου. Λοιπόν, Κοιτάξτε, κοιτάγατε τις καμπίνες, έχουμε τρεις διερμηνείς ανά καμπίνα. Αυτή είναι η έκφραση. Με καταλαβαίνετε. Να σας απαντήσω στα ισπανικά. Οπότε ε, προς τούτο βάλτε τα ακουστικά και, έτσι θα εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν από την διερμηνία αυτή η δυνατότητα του κανείς μπορεί να μιλά τη μητρική του γλώσσα για να μπορεί έτσι ορθά να τοποθετηθεί σε σχέση με όσε σκέψεις έχει και να μπορεί να περάσει αυτό το μήνυμα για όλους. Όλοι επομένω να μπορούν να ε, ε, εκφραστούν και να ε, ε, κατανοήσουν τις γλώσσες. Αυτό είναι κάτι το οποίο ορίζει το πρώτο άρθρο της Ρώμας που λέει ότι υπάρχει ίση μεταχείριση, υπάρχει μεταξύ των γλωσσών και ότι πρόκειται για ένα δικαίωμα το οποίο δεν μπορεί να απεμποληθεί το δικαίωμα χρήσης της μητρικής γλώσσας και οπότε είτε μα αρέσει είτε όχι πρόκειται επομένω για θεσμικού και συνταγματικού χαρακτήρα δέσμευση. Και πρόκειται επομένω για κάτι ε, το οποίο αποφασίστηκε με την ομοφωνία όλων των κρατών μελών. Οπότε, όσο και να μας αρέσει να αναπτύσσουμε επιχειρήματα, πρόκειται επομένω για ζήτημα πολιτιστικό, πολιτικό, ε, ουσιαστικά ηθικό. Και οπότε ε, θα πρέπει αυτό το ζήτημα να συζητηθεί. Τώρα στα γαλλικά, εάν ρωτήσετε πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να υπάρχει κάποια εξοικονόμηση δαπανών και πώς τα θεσμικά όργανα μπόρεσαν επίσης να συμμετάσχουν σε αυτή την συλλογική προσπάθεια θα σας έλεγα ότι είμαι υπάλληλο και οι, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έκαναν ακριβώς αυτό που έκαναν και τα κράτη-μέλη περιέκοψαν προσωπικό. Έχουμε μια σημαντική συρρήγνωση ε, στο οργανόγραμμα για να αναλύσουν τα πέντε αιτίες. Έχουμε ε, αναθεωρήσει την διαδρομή των σταδιοδρομιών, ούτως ώστε ε, να έχουν περικοπεί οι προαγωγές, έχουμε αναδιαρθρώσει βάθρων την οργάνωση των υπηρεσιών μας, οπότε και εμείς οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκή Ένωσης βάζουμε το λιθαράκι μας στον εξορθολογισμό της χρήσης των πόρων. Και οπότε θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, με το πώς λειτουργούν τα εθνικά κοινοβούλια. Αν κάναμε αυτή τη σύγκριση θα διαπιστώναμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι Ευρωβουλευτές έχουν αρμοδιότητες, έχουν ευθύνες πιο μεγάλες από αυτό που πρώτης όποιος κανείς ε, νομίζει. Οπότε αυτό έχει να κάνει και με το ότι ένας Ευρωβουλευτής και προσωπεί πολύ περισσότερους Ευρωπαίους από ότι ένας Εθνικός Βουλευτής. Οπότε και εδώ νομοθετούμε για 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους σε 24 γλώσσες, οπότε αυτό το νομοθετικό έργο αντιστοιχεί στο 80% των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Οπότε αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αποτελεσματικό, διακρίνεται από διαφάνεια και επίσης θέτει στην διάθεση του Ευρωπαϊκού Πολίτη πληροφορίες, ενημέρωση και μέσα ε, συμμετοχής σε αυτό το γίγνεσθε που δεν ισχύει το ίδιο για τα εθνικά κοινοβουλία. Και αυτό σας το λέω κατηγορηματικά. Σας το λέω με βεβαιότητα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθουμε περήφανοι για το έργο το οποίο επιτελούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρόκειται απλώ εδώ για μια διασπάθηση χρημάτων. Δεν πάει να πει αυτό Ευρώπη. Μπορούμε να βελτιωθούμε και βεβαίω θα πρέπει να έχουμε βίκονους προ προς αυτούς που απευθύνονται προς εμάς, οπότε μπορούμε να τα καταφέρουμε και ο Γενικό ε, γραμματέα δεν θα διαψεύσει τις ε, διαβεβαιώσει που σα παρέχω. Πρόκειται για μια διαδρομή, δύσκολη βέβαια, ε, αλλά αν θέλουμε θα τα καταφέρουμε. Αυτό είναι το μήνυμα ε, το, το οποίο έχουν όταν ακούει να ακούει Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτές οι περικοπές, αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυστηρότεροι από τους αντιστοίχους εθνικούς ελέγχους. Υπάρχουν αυτές τις διαδικασίες ελέγχου που αφορούν και το τελευταίο ευρώ. Γιατί πρόκειται εδώ για τον ε, δημόσιο κορβανά, για δημόσιο χρήμα. Όλα διέπονται από διαφάνεια. Α, ναι, Δανέσκα θα ήθελα να μπορώ να σας μιλήσω, αλλά δεν γνωρίζω. Ευχαριστώ πολύ, <coughs> κύριε Λάους. θα πρέπει να αντικαταστήσω λιγάκι τον κύριο Κλάους Βέλε μάλλον θα πρέπει να δώσω το λόγο στον κύριο Κλάου Ρέλε, ο οποίο ήρθε και ο οποίος θα σα ε, παρουσιάσει τώρα τι κύριε πολιτικέ γραμμέ. Καταρχήν σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο τη συνθήκη τη Λισαβόνα στη διαδικασία εκλογής του Πρόεδρου της Κομισιόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Πώ τα πράγματα έχουν αλλάξει, πώ έχει υπάρξει μια αλλαγή η οποία επηρέασε και την εκλογική εκστρατεία. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Πάουλγερ, από την Κομισιόν για την παρουσία του και για την πλήρη συνεργασία του τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες. Καλημέρα σας, λέει ο κύριος ε, Κλάους Βέλε. Όπως ξέρετε, έχουμε επιλέξει ένα φιλόδοξο τίτλο για την εκστρατεία μας, που λέγεται αυτή τη φορά είναι αλλιώ. Μια μεγάλη πρόκληση βεβαίως ε, ένα τέτοιο αποτέλεσμα αλλά θεωρούμε πως έχουμε ε, επαρκείς λόγους για να λέμε κάτι τέτοιο. Πολιτικά συνέβησαν πολλά πράγματα τα τελευταία πέντε χρόνια που αφορούν τους πολίτες πολύ πιο άμεσα από ό,τι στο παρελθόν. Ειδικά από την οικονομική κρίση τα μέτρα στις χώρες ε, που είναι σε πρόγραμμα οδήγησαν σε κάποια μέτρα τα οποία λαμβανόταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επηρέαζαν άμεσα τις κοινωνικές και οικονομικές ε, συνθήκες. Αλλά εγώ θα έλεγα πως αυτό ισχύει και σε άλλες χώρες που γλίτωσαν αυτή την ε, μοίρα, αλλά έπρεπε να λάβουν μέτρα, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, αλλά και οι χώρες που έλαβαν κάποιες ε, δημοσιονομικές εγγυήσει, γιατί οι πολίτες αντιλήφθησαν πως οι εγγύησει αυτές ήταν τεράστιες και όταν δίνει κανείς εγγυήσεις δεν μπορεί να αποκλείσει μία μέρα να χρειαστεί να καταβληθούν αυτές. Οπότε η δημοσιονομική χρήση, το χρέος, όλα αυτά οδήγησαν τον κόσμο να καταλάβει πως οι αποφάσεις σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο αφορούν τον πυρήνα των συνθήκων των οικονομικών που ζουν. Επίσης νομικά ε, έχουμε μια αλλαγή. Η συνθήκη της Λισαβόνας επέθυνε ισχύει την 1η Δεκεμβρίου 2009. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι έγινε αφού ανέλαβε καθήκοντα η Ευρωπαϊκή σημαινει οτι είναι αφου ανελαβε Οπότε τα κομμάτια εκείνα που αφορούν τον ε, διορισμό Προέδρου και της Κομισιόν ολόκληρης ε, δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα. Οπότε είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται η συνθήκη της Λισαβόνας ως προς αυτό. Και σε τι διαφέρει. Σε τρία πράγματα. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν κάνει πρόταση για πρόεδρο της Κομισιόν ε, πρέπει να λάβει υπόψη το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Βεβαίω, η όλη συζήτηση μετά είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, πώς το μετράμε, αλλά το σαφές είναι πώς ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη από το Συμβούλιο. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι πλέον κομμάτι της συνθήκης δεύτερον. Μετά τις ευρωεκλογές πρέπει να υπάρξει μια διαβούλευση του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι στην δήλωση υπαρθμών 11 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Οπότε πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα συνεννόησης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δει και ο πρόεδρος του Συμβουλίου το πώς θα λειτουργήσει η υπόθεση αυτή. Και η τρίτη αλλαγή είναι μια πάρα πολύ σημαντική διευκρίνηση. Η διευκρίνηση αυτή είναι πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο της Κομισιόν. Η διατύπωση πλέον δεν είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει, εγκρίνει. Η διατύπωση είναι εκλέγει. Οπότε, η πραγματική απόφαση θα ληφθεί όταν εκλέξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόεδρο της Κομισιόν. Αυτά τα τρία στοιχεία δεν υπήρχαν. Οπότε όλα αυτά μαζί δημιουργούν μια νέα κατάσταση νομική. βεβαίω δεν απαντάνε σε όλα τα διαδικαστικά ζητήματα, γι' αυτό ακριβώς ε, τα συζητάμε αυτά δημοσίως και με τις κυβερνήσεις, το τι θα γίνει ακριβώς και τι σημαίνουν αυτά ακριβώς, αλλά η πρόθεση της συνθήκης της Λισαβόνας είναι σαφώς να ενισχυθεί η συνεισφορά του εκλογικού σώματος ε, και του Κοινοβουλίου ως ε, θεσμικό όργανο. Ε, με βάση αυτά τώρα για πρώτη φορά όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμματα έχουν αποφασίσει να υποβάλουν κάποιες υποψηφιότητες. Ε, τι σημαίνει λοιπόν λένε τώρα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Σημαίνει πως πρέπει να υπάρχει πολύ πιο στενή σχέση μεταξύ προεκλογικής εκστρατείας ε, πολιτικών πλειοψηφιών και δεν θα σας πούμε μόνο εκ των υστέρων του τι σημαίνει η νέα διαχείριση της ε, Κομισιόν αλλά θέλουμε να πούμε εκ των προτέρων ποιοι είναι οι υποψηφοί μας και εμφανίζονται δημοσίως ε, στην τηλεόραση, στα ΜΜΕ γενικώ ε, για να είναι γνωστές οι επιλογές πριν ε, από το αποτέλεσμα. Και βεβαίως έχουμε και κάποια προσωποποίηση αν θέλετε της εκστρατείας αυτής. Γιατί αν το δείτε και σε εθνικό επίπεδο, εάν οι εκλογές ήταν μόνο για την σύνθεση του Κοινοβουλίου και δεν είχαν ούτε μία σχέση με την κυβέρνηση, με την εκτελεστική εξουσία, οπωσδήποτε θα ήταν πολύ χαμηλότερο το ενδιαφέρον του κοινού και η προσέλευση. Υπήρχε αν ψήφιζαν για τη Γερμανική Βουλή μόνο οι Γερμανοί, ε,

Δεν έχει καμία σύγκριση με το τι γινόταν πέντε χρόνια πριν. Και μπαίνουμε στην τελευταία φάση πλέον τη εκστρατεία όπου θα παίξει σημαντικό ρόλο η τηλεόραση. Τέλο, λίγα λόγια για την διαδικασία που θα ακολουθήσει. Όπω ξέρετε, μέχρι, τις, μέχρι και τι 25 έχουμε εκλογέ. Αλλά ήδη από την Πέμπτη θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε κάποια νούμερα, αποτελέσματα, δημοσκοπήσεις ε, θα τα κάνουμε πιο εύκολα, πιο ευανάγνωστα με το να τα μεταφράζουμε σε έδρες ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, ε, δεν το είχαμε κάνει στο παρελθόν. Και αυτό το κάνουμε γιατί βεβαίως χρειάζεται εξειδίκευση να το κάνει κανείς για 28 χώρες και δεν είναι καθόλου εύκολο. Και επιτρέπει ευκολότερα να αντιληφθεί κανείς το τι διακυβεύεται τι μπορεί να αναμένει κανείς, ε, ποια είναι η πραγματική αύξηση της ε, άκρας δεξιάς, ε, της πολύ αριστεράς κτλ. Οπότε και βεβαίως το βράδυ των εκλογών, τα βράδια των εκλογών θα προσπαθήσουμε να σας δίνουμε πληροφορίες και το τι συμβαίνει σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις και όταν κλείσουν οι τελευταίες κάλπες 11 η ώρα το βράδυ στην Ιταλία θα έχουμε πολύ συγκεκριμένα νούμερα για το πώς θεωρούμε ότι θα έχει η νέα σύσταση του Κοινοβουλίου και βεβαίως με το ποσοστό αβεβαιότητας το οποίο είναι πολύ υψηλότερο στις 11 από ότι μία και 2 και 3 ώρες μετά Νομίζω πως ε, καλύτερο είναι να κάνουμε μια τέτοια πρόβλεψη, να σας δώσουμε ένα πιο ακριβές νούμερο. Μετά, πολιτικά, στις 27 Μαΐου θα συναντηθούν ε, όλοι οι επικεφαλείς ε, των πολιτικών ομάδων με τον Πρόεδρο. Στις 27 το απόγευμα θα έχουμε την διάσκεψη κορυφής των διαφόρων πολιτικών οικογενειών και 27 το βράδυ το άτυπο δείπνο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα προσπαθήσει επίσης να ερμηνεύσει την κατάσταση και να δώσει ίσως μία εντολή στο Χέρμαν Φανρομπάι για το τι μπορεί να κάνει και ίσως να δώσει και κάποιες πολιτικές ενδείξεις. Μετά οι πολιτικές ομάδες ε, θα συνέλθουν σε σώμα. Αυτό μέχρι τις 18 Ιουνίου, οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι θα είναι τελευταίες ομάδες, οπότε 18 Ιουνίου όλες οι ομάδες έχουν συνέλθει με νέες ηγεσίε, θα έχουν συσταθεί σε σώμα και το αργότερο στις 24 Ιουνίου όλες οι ομάδες πρέπει να αποστείλουν την τελική τους σύνθεση κάτι το οποίο βεβαίως έχει μετά τη σημασία για το ποιες θέσεις θα καταλάβουν οπότε αυτά θα οριστικοποιηθούν στις 24 γιατί βεβαίως όλοι θέλουν να έχουν τους μεγαλύτερους αριθμούς και αυτό τρεις μέρες πριν από τις 27 Ιουνίου όταν θα συνέλθει επισήμως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα κάνει μια πρόταση για πρόεδρο της Κομισιόν μετά 1η Ιουλίου θα εκλεγεί και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις 16 Ιουλίου αν δεν κάνω λάθος ε, ε, είναι η πρώτη δυνατότητα να εκλεγεί η πρόεδρος της Κομισιόν βεβαίως αυτή είναι η καλύτερη περίπτωση το πιο αισιόδοξο σενάριο αλλά βεβαίως και στο παρελθόν είχαμε εκλογή πρόεδρο της Κομισιόν το Σεπτέμβριο, κάτι το οποίο βεβαίως μετά είχε ως αποτέλεσμα και άλλες καθυστερήσεις για την στελέχωση ολόκληρης της Κομισιόν. Ελπίζω λοιπόν να ήταν ε, σαφής και επαρκής αυτή η εισαγωγή. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, έχετε το λόγο τώρα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Έρχομαι από την Ελλάδα. είδα ότι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την ε, νέα κατάσταση ότι θα εκλεγεί ο πρόεδρος της Κομισιόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φοβάμαι όμως ότι υπάρχουν πολλοί αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν εκλέγονται. Ο κύριος Φανρόμπα, η κυρία Άστον, παραδείγματος χάρη, δεν έχουν εκλεγεί από κάποιον. Ποιο θα του εκλέγει λοιπόν, σε ποιον είναι υπόλογοι και το ίδιο ισχύει και για του επιτρόπου. Δηλαδή, δίνεται πολύ έμφαση στην εκλογή μονάχα ενό αξιωματούχου. Αυτό οδηγεί σε μια χαλαρότητα και ουσιαστικά οδηγεί σε αποξένωση των πολιτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν φτάνει ένα. Ναι, το ερώτημά σα είναι ποιο έχει επιλέξει και την κυρία Άστον και τους επιτρόπους, μα το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο τους έχει εκλέξει γίνεται μια ψηφοφορία στο τέλος της διαδικασίας όπου γίνεται η επίσημη εκλογή τους ως συλλογικό σώμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προηγούνται ακροάσεις και το αποτέλεσμα των ακροάσεων πολλές φορές ήταν ότι ορισμένοι μεμονωμένοι υποψήφοι, εάν θεωρηθούν ότι δεν είναι αρκετά επαρκείς, αποσύρονται. Αυτό δεν το βλέπετε σε εθνικό επίπεδο με υπουργού. Πολύ σπάνια μπορεί ένα κοινοβούλιο να εξασφαλίσει ότι θα, δεν θα γίνουν δεκτοί ορισμένοι ω υπουργοί σε μια κυβέρνηση. Σίγουρα η εντολή που έχουμε οι, η επίτροποι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο <clears throat> δεν είναι πιο αδύναμη από την εντολή που έχουν οι, οι υπουργοί στα Εθνικά Κοινοβούλια. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι υπουργοί πρέπει να είναι βουλευτές, σε άλλες περιπτώσεις όχι. Ο κύριος Φαν Ρομπόι έχει επιλεγεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Αν θέλετε να τον εκλέξουμε εμείς αυτό θα μας άρεσε βέβαια. Εάν προτείνετε να εκλέγετε από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θα ήταν ένα ακόμα πιο επαναστατικό σενάριο, αλλά σίγουρα έχει μια εντολή που απορρέει από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπετε πολλές φορές να γράφει ο Βρετανικός τύπος ότι δεν έχουν εκλεγεί όλοι αυτοί είναι εξίσου εκλεγμένοι με πολλούς από τους αξιωματούχους της Βρετανικής κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ από την Σλοβάκια Πράγοντα για την προεκλογική εξαρτία. Πολύ καλό είναι να έχουμε υποψηφίους για την Προεδρία της Κομισιόν και αυτό κάνει πιο απλή τη δουλειά του δημοσιογράφου, γιατί προσωπικοποιείται η προεκλογική εκστατεία μεταξύ του Σούλτς, του Γιούνκερ, του Τζίπρα, της Κέρα κτλ. Από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ξέρετε κάποιον, κάποιον από τους φίλους σας, ίσως ο οποίος θα ψήφιζε για τους συντηρητικούς ή για τους σοσιαλιστές ή για κάποιον άλλο, γιατί ξαφνικά έχουν εμφανιστεί κάποιοι υποψήφοι. Δεν ξέρω κάποιον Σλοβάκο ο οποίος θα ψήφισε τους Σλοβάκους σοσιαλδημοκράτες γιατί απλώς είναι υποψήφιος ο κύριος Σούλτς. Αν δεν είναι ρητορικό ερώτημα ή πραγματικό ερώτημα, ναι, ξέρω πολλούς οι οποίοι θα <clears throat> ενδιαφερθούν λόγω των υποψηφίων που παρουσιάζονται. Είναι πολλοί στο βελίο οι οποίοι αναρωτιούνται ποιο βελικό κόμμα θα πρέπει να ψηφίσουν για να υποστηρίξουν ένα, δεδομένο επικεφαλής υποψήφιο. Ξέρω από το προσωπικό μου κύκλο, αλλά αυτό μπορεί να είναι μονάχα προσωπικό μου θέμα, ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το ποια κόμματα σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να υποστηριχθούν στις ευρωεκλογέ για να υπάρξει το σωστό αποτέλεσμα σε σχέση με τον πρόεδρο της Επιτροπής. Αυτό μπορεί να είναι, αν θέλετε, μια ειδική περίπτωση. Αλλά εγώ βλέπω στο δικό μου στενό κύκλο να υπάρχει μια μετατόπιση από την παραδοσιακή ε, εκλογική συμπεριφορά. Υπάρχει ένας νέος τρόπος απόφασης για το ποιο κόμμα θα ψηφίσουν λόγω της δυνατότητα εκλογής του Προέδρου της Κομισιόν. Δεν λέω ότι αυτό συμβαίνει σε όλους, αλλά πιστεύω ότι κάποιοι μπορεί να επιχειρηματολογούν με αυτόν τον τρόπο, ιδίως μετά τις ε, συζητήσεις, τα debates στην τηλεόραση λένε πώς θα εξασφαλίσω ότι ο Α και όχι ο Β θα γίνει πρόεδρος της Κομισιόν. Αυτό μπορεί να διαφοροποιήσει λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο ψηφίσουν οι εκλογείς. Έχουν μία γραμμή για τις εθνικές εκλογές και μία διαφορετική γραμμή λοιπόν για τις ευρωεκλογές ενδεχομένως. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Από το Ελπεριόδικο καταλούνια για τις αλλαγές οι οποίες έχουν εισαχθεί από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτές οι αλλαγές είναι βέβαια ένα μεγάλο βήμα, όπως είπε και ο συναδελφός μου, αλλά είναι κάπως ασαφής. Για να επανέλθω σε αυτό που είπατε, είπατε ότι η Κομισιό πρέπει να λάβει υπόψη τις τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Να λάβει υπόψη, αυτό όμως δεν είναι ακριβώς σαφές, και στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα κάνει κάποιες διαβουλεύσεις για το θέμα αυτό. Όλα αυτά είναι κάπως ασαφή πώς μπορούν αυτές οι αλλαγές να τροποποιήσουν την ισορροπία δυνάμεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν είναι τόσο περιορισμένες. Νομίζω ότι η απάντηση είναι ότι είναι η πρώτη φορά, είναι το πρώτο παράδειγμα μια τέτοια εκλογή που θα δημιουργήσει και κάποιο προηγούμενο. Νομίζω ότι πολλά εξαρτώνται από το τι θα γίνει τώρα. Αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, παραδείγματο χάρη, αποφασίσει να ματαιώσει αυτή τη διαδικασία και να μην ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών όταν οι επικεφαλείς υποψήφοι έχουν εμφανιστεί σε debate, στην τηλεόραση, σε δημόσιες συγκεντρώσεις. Αυτό δίνει την προσδοκία στους πολίτες ότι θα παίξει κάποιο ρόλο η δική τους ψήφος σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βέβαια να ακολουθήσει μία άλλη γραμμή. Αυτό θα ματαιώσει τις προσδοκίες των πολιτών και μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Επομένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτό το ενδεχόμενο. Όλα εξαρτώνται από το πώ θα λειτουργήσει αυτή η διαδικασία την πρώτη φορά που εφαρμόζεται, κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δέχεται αυτή τη λογική ή την απορρίπτει και δεύτερον, δεχόμαστε εμείς τη λογική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Γιατί οι πραγματικές εκλογές λαμβάνουν χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμφωνεί, δεν είναι υποχρεωμένο να δώσει 376 ψήφου στον υποψήφιο που προκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τότε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να επανέλθει σε ένα μήνα με ένα νέο υποψήφιο. Επομένω δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε απόλυτα με τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τόμα Άιφερτ από την ε, Wiener Zeitung. Μία τεχνική ερώτηση. Τι προτείνετε σε εμά ω ε, δημοσιογράφου για την κάλυψη των εκλογών στι 25 Μαου. Είπατε στι 11 11 η ώρα κλείνουν οι κάλπες στην, Ιταλία. Ξέρουμε από τα προηγούμενα παραδείγματα, από προηγούμενες εκλογές, ότι θα έχουν μέχρι τότε διαρρεύσει κάποια αποτελέσματα. Αν εσείς ήσασταν στη θέση μου, στο γραφείο μου, την Κυριακή το βράδυ, τι θα κάνατε. Πώς θα σχεδιάζετε την μετάδοση των αποτελεσμάτων και τον σχολιασμό τους. Ναι. νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν παρουσιάσει βοηθούν γιατί από τον Σεπτέμβριο έχουν γίνει κάποιες κινήσεις αλλά περιορισμένου βεληνικούς οπότε ε, θα πρέπει να αποφύγουμε τα ακραία σενάρια. Για να λέμε ότι έχουμε 250 μέλη τα οποία θα ανήκουν στα άκρα γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει το κοινοβούλιο. Υπάρχουν τα στοιχεία αυτά επί τη βάση ε, του ΖΕΝΕΣ που είναι φορέας ε, επαγγελματικό με τη Γαλλία και αυτό που θα ήθελα να συμβουλεύσω για το βράδυ των εκλογών είναι το ότι αν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ε, από σκοτεινή πηγή και που κατατείνουν το αντίθετο από το αναμενόμενο, θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός. Επίσης, προετοιμαζόμαστε ούτως ώστε την εκλογή βραδιά να σας δώσουμε και πληροφορίες για κάποια θέματα κλειδιά. Αυτά που θα κάνουν την εργασία εδώ πιο ελκυστική. Ας πούμε, background για κάποια ζητήματα. Κλειδιά τι είναι. ότι αν υπάρξει κάποια καινούργια πολιτική ομάδα της ε, άκρας δεξιάς, βεβαίως και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, εάν υπάρχουν πολιτικές ομάδες θα μπορούσαν να ξαναμπούν στο κοινοβούλιο και αυτό βεβαίως είναι ενδιαφέρον θέμα και επίσης έχουμε και κάποιες προκλήσεις δηλαδή ατομικές προσέξεων ενδιαφέρον ας πούμε ο, ο Μάρτιν Κελέναν ε, των συντηρητικών θα δώσει σκληρή μάχη στην εκλογή του περιφέρεια και δεν είναι βέβαιο να τα καταφέρει να επανεκλεγεί. Οπότε και σε σχέση με αυτή την προσπάθεια επανεκλογής θα σας ενημερώνουμε για το κατά πόσο θα καταφέρει ή όχι. Και τι θα γίνει με την πολιτική ομάδα, ας πούμε, των 40, 50, 60 μελών, αν τον έχει ηγέτη. Όλα αυτά επομένω, τα, τα, τα επιμέρου ζητήματα μέχρι ότου έχετε την ενημέρωση για τα γενικότερα. Θέματα λοιπόν προσφέρουν ενδιαφέρον για τους αναγνώστες σας. Ε, μία δεύτερη ερώτηση, συγγνώμη. Περιμένετε κάποια αποτελέσματα ή κάποια καταρχήν αποτελέσματα να βγουν πιο νωρίς, ε, ε, και μετά να έχετε τα υπόλοιπα στις 5-6 το απόγευμα συμπληρωματικά. Ναι, ναι, είναι πολύ πιθανό λέει ο Γενικός Γραμματέας. Ήδη με τις προπάρχουσες πληροφορίες μπορείτε να έχετε αυτά σαν μπούσουλα για να δείτε ακριβώς ε, τι γίνεται σε περίπτωση που δεν μπορείτε να επαληθεύσετε κάποιες πληροφορίες και οπότε να μπορείτε να βασίσετε σε αυτά τα στοιχεία για να κάνετε ένα ρεπορτάζ. Άλλες δύο ερωτήσεις. Εσείς, η κυρία, θέλετε το λόγο να. Εσείς πρώτα. Γι' αυτό για την αλλαγή των συνθήκων είναι θέμα. Και επίσης η ερμηνεία για το αποτέλεσμα των εκλογών, όπως μας τα είπατε, είναι ερμηνεία του τι ισχύει στην Ευρώπη και στο Κοινοβούλιο, αλλά όχι στην Επιτροπή. Γιατί, όπως είπατε προηγουμένως, η επικοινωνία μετά τις εκλογές θα αφορά κυρίως το κατά πόσον τα κρατημέλη με το Συμβούλιο αν θα μπορέσουν πώς να το πω κατά πόσον θα παίξουν το παιχνίδι ή δεν θα παίξουν το παιχνίδι το οποίο προσδοκάται γιατί αυτό θα έχει σχέση με το κατά πόσον έχει ψηφιστεί ο πρόεδρος που ήθελαν ή όχι. Υποθετική είναι η ερώτηση, αλλά είναι και κάτι άλλο. Έχετε κάποιο feedback από κομισιόν, από ε, κράτη-μέλη για το τι στάση θα υιοθετήσουν μετά τις εκλογές. Γιατί ήδη κυκλοφορούν κάποιες απόψεις ότι έχουμε ε, κάποια τέτοιου είδους χειραγώγηση που θα αυξήσει την δύναμη του Κοινοβουλίου. Κάτι σαν απειλή. Ναι, ναι, αυτό όμω δεν είναι το χειρότερο. Περισσότερη δημοκρατία είναι το θέμα, Λέω ο εσεί Εσείς, λέγω με Μούλερ, από τη ρυθμίδα Ελμούντο τη Μαδρίτη. Θέλω να μιλήσω ισπανικά. Θεωρώ ότι αυτή η ερώτηση αυτό της συναδέλφου ε, από την εφημερίδα El Periódico. Είναι το σημείο κλειδί για την επίσκεψή μας, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολύ διφορούμενο αυτό που λέει η συνθήκη σε σχέση με τις ε, εκλογές αυτές. Ε, εμείς που υπέστημεν την εισβολή του Ναπολέοντα, έχουμε κάποια προβλήματα, ούτω ώστε το εθνικό δίκαιο να το χωνέψουμε. Τι θα γίνει τα πράγματα, θα συνήθω ισχύουν ακριβώ όπω έχουν σήμερα. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε αυτά να τα θεωρήσουμε μια πραγματικότητα που θα την καταπιούν, που την χωνέψουν οι συμπολίτε μα. Και όπω είπε ε, μια συνάδελφος, υπάρχει κάποιο είδου μπούσουλα, κάποιο είδου χάρτη πορείας που έχει το κοινοβούλιο, ούτω ώστε κάποιο θα πρέπει τελικά να, να αναδιαπιστώσει κατά πόσον αυτά που πιστεύετε είναι αυτά που λένε οι συνθήκες. Υπάρχει τέλος πάντων κάποιο είδους τρόπος να επιλύσουμε, να βρούμε τη διέξοδο ε, από αυτό το διέξοδο, από αυτή την, την σύγκρουση. Γιατί έχουμε αυτούς τους ε, υποψήφιους για Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι κάποια πρόσωπα που ούτε καν κατεβαίνουν σε εκλογές. Uh, I, think first it's very... Νομίζω πως πρώτα απ' όλα πρέπει να θυμόμαστε πως εκεί αυτοί οι υποψηφοί δεν έχουν προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καμιά φορά υπάρχει αυτή η εντύπωση. Ε, δεν συμβαίνει αυτό όμως. Αυτό το κάνει το, κάθε κόμμα το οικείο κόμμα. Ποια είναι αυτά τα πολιτικά κόμματα, μα αποτελούνται από τα εθνικά κόμματα, τους ηγέτες τους, τους αρχηγούς κατών και κυβερνήσεων. Μπορείτε να είστε σίγουροι πως ούτε στο ΕΛΚΑ, ούτε στους σοσιαλιστές, ούτε στους φιλελεύθερους ε, θα μπορούσε να έχει οριστεί κάποιος ως υποψήφιος για πρόεδρος της χωρίς την έγκριση όλων των ε, πρωθυπουργών ε, ή τουλάχιστον πάνω από 90% όσων βρίσκονται γύρω από το τραπέζι. Αντιθέτως, ε, έχουν εμπλακεί πάρα πολύ στις υποψηφιότητες αυτές. Οπότε θα είναι λίγο περίεργο μετά να πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να μην τον ξέρουν τον άνθρωπο αυτόν. Γιατί έχουν οριστεί, όπως είπα, από τα ε, ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα με την στήριξη των Πρωθυπουργών. Δεν μπορεί μετά να πάνε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να τους πούνε δεν σε ξέρω, δεν σε είδα. Δεν είναι και πολύ πιστικό. Μπορεί κάποιος να έχει επιφυλάξεις για τον υποψήφιο άλλου κόμματος, να πει ότι δεν τον έχει δει, αλλά τουλάχιστον οι 12-13 πρωθυπουργοί του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ξέρουν τον υποψηφιό τους, τον έχουν υποστηρίξει. Και οι άλλοι 12-13 των σοσιαλιστών. Το ίδιο. Δεν είναι λοιπόν οι υποψήφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι των Ευρωπαϊκών Κομμάτων με την πλήρη στήριξη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Είναι σαφές. Δεν μπορεί να πει μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν τους ξέρουμε και δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Βεβαίως ε, το κάθε κόμμα είναι μειοψηφία, οπότε το ζήτημα είναι μετά πώς περνάμε από την μειοψηφία στην πλειοψηφία υποψήφιος του ΕΛΚ ε, δεν θα έχει πλειοψηφία ούτε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ούτε στο Κοινοβούλιο το ίδιο και ο Σοσιαλιστής μόνο το δικό του κόμμα οπότε εκεί θα ξεκινήσει η πολιτική συζήτηση αλλά η εντύπωση που δημιουργείται ειδικά από τους συμβούλους πως οι άνθρωποι αυτοί είναι άγνωστοι και εμφανίστηκαν από το πουθενά είναι παράλογη η περιγραφή της κατάστασης. Και νομίζω έτσι απάντησαν μέρη και στην άλλη ερώτηση. Οπότε δεν είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται από το πουθενά έχουν οριστεί ως υποψήφοι με μια διαδικασία με τη στήριξη των αρχηγών κρατών κυβερνήσεων. Το ζήτημα είναι πώς περνάμε από την μειοψηφία, γιατί ακόμα και το μεγαλύτερο κόμμα θα είναι μειοψηφία, σε πλειοψηφία. Χρειάζεται ειδική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ειδική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι ακριβώς η ίδια, η οποία βέβαια σημαίνει πως πρέπει να υπάρξουν πολιτικές συμμαχίες. Αυτό ακριβώς ψάχνουμε. Τώρα έχουμε μια νέα ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ναι, γιατί έχουμε νέα συνθήκη. Κάποιοι είχαν ξεχάσει τη συνθήκη της Λισαβόνας γιατί έχουν περάσει πέντε χρόνια, αλλά υπάρχει η συνθήκη της ε, Λισαβόνας. 28 κράτη-μέλη, 28 εθνικά κοινοβούλια την ενέκριναν ε, και ακριβώς ε, θα γίνει πιο αποφασιστικό ο ρόλος των ευρωεκλογών και για την εκλογή της ε, Κομισιόν και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βέλε, κύριε Λούς. Με συγχωρείτε. Μία γρήγορη ερώτηση αν μπορώ να κάνω από το Λουξεμβούργο Βολφαν Λάιτσιχ. Έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου όσο περνά ο χρόνος, αλλά η προσέλευση στις ευρωεκλογές ε, διαρκώ. Ε, μειώνεται. Δεν σας ανησυχεί αυτό, δηλαδή, εάν ε, για ακόμη μια φορά έχουμε μειωμένη προσέλευση, δεν ε, υπονομεύεται έτσι η δημοκρατική νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τι προσέλευση αναμένετε εσείς. Ναι, κοιτάξτε για την προσέλευση. Η προσέλευση από το 1979 κινείται παράλληλα με την προσέλευση στις εθνικές εκλογές, δηλαδή έχει πτωτική τάση. Αλλά δεν είναι πιο χαμηλά από τις εθνικές εκλογές. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία, ξεκινώντας από χαμηλότερη αφετηρία. Και αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι πως ε, η αφετηρία αυτή η χαμηλότερη ήταν ε, λόγω του ότι εδώ πέρα αποφασίζουμε μόνο, είχαμε μάλλον, την απόφαση μόνο για την σύνθεση του Κοινοβουλίου και όχι για το ποιος θα είναι η κυβέρνηση. Αν λοιπόν βγάζαμε και στις Εθνικές Βουλές το αντίστοιχο, δηλαδή μόνο την ομοθετική και όχι την εκτελεστική εξουσία, προφανώς και εκεί πέρα η προσέλευση στο εθνικό επίπεδο θα ήταν πολύ χαμηλότερη. Αυτό είναι βασικό επιχείρημα ε, για εμάς για να πούμε πως πρέπει να συνδεθεί η σύσταση, η σύνθεση του Κοινοβουλίου με το ποιος ασκεί την εκτελεστική εξουσία. Δεν μπορεί να μην φανεί τώρα, αλλά σε μία, δύο, τρεις εκλογικές αναμετρήσεις νομίζω θα είναι σημαντική η επίδραση. Οι ενδείξεις που έχουμε τώρα είναι πως αυτοί που είναι αποφασισμένοι να ψηφίσουν σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από 5 χρόνια είναι κατά 3% περισσότεροι. Δεδομένου του ότι από το 1979 ε, είχαμε συνεχώς πτωτική τάση, εάν μπορούμε να σταθεροποιήσουμε την προσέλευση ή και να έχουμε μία μικρή αύξηση, αλλά αυτό το ξέρουμε μόνο στις 25 Μαΐου, ε, νομίζω πως θα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα, όντως. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάλι όλους σας. Θα διακόψουμε για 10 λεπτά. Για... Σας παρακαλώ να επανέλθετε.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 avons abordé cette élection avec beaucoup de respect, car nous avons tous été admiratifs de la façon dont les Tunisiens ont conduit leur révolution. Supporting the process of change too, as we've described in Tunisia and Egypt, Libya and Yemen, other countries of the Middle East and North Africa, requires our continued support for the first time in a long time as the international community uniting towards an action on Syria.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 They think the European Union is their enemy. And indeed it is. Et je suis convaincu que si l'Europe succombe aux sirènes populistes et eurosceptiques, nous remonterons le fil du temps en sens inverse. Ce serait un retour vers le chaos et la guerre pour l'Europe. And only a strong and united Europe can defend our interests globally from labor rights to climate change. After the European wars, we owe a lot to the rest of the world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 adopted. Acuerdo comercial de lucha contra la falsificación y el acuerdo ha sido rechazado. If we think about these systems as a whole, we actually have a planetary surveillance system that is not accountable to the people, that is used for extrajudicial assassination. Nous passons au dossier SWIFT en raison de la surveillance exercée par la NSA.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 Congratulazioni onorevole Tremosa. The ECB must ensure that in the exercise of its responsibilities there is the highest degree of transparency and accountability. The very high bonuses that are still being paid to bankers suggest that there are excessive profits in the banking sector. Les conséquences économiques et sociales graves que connaissent aujourd'hui certains États membres auraient pu être évitées, ce qui sera corrigé maintenant par la combinaison du six pack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 that the signatories to the intergovernmental agreement on the transfer and mutualisation of Contribution to the single resolution fund are ready to declare that they will strive to complete its process of ratification in accordance with their respective national legal requirements. l'union bancaire c'est clairement la pierre centrale. nous avons mis de la transparence de la responsabilité j'ose prononcer à nouveau le mot de morale et d'éthique là où elles avaient disparu.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 Okay, so your attention, please. Θα ήθελα να έχω την προσοχή σας παρακαλώ. Καθίστε παρακαλώ. Συνεχίζουμε με το δεύτερο τμήμα του σεμιναρίου μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να καλωσορίσω στο σεμινάριό μας την κυρία Ποδηματά. Η κυρία Ποδηματά είναι ευρωβουλευτής από την Ελλάδα είναι στο Σοσιοδημοκρατικό Κόμμα και είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αρμόδια για τα θέματα επικοινωνίας στο Προεδρείο. Η κυρία Ποδηματά είναι και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και ως μέλος αυτής της Επιτροπής έχει συντάξει μια πολύ σημαντική έκθεση για την φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. έχει, είναι απόφυτος της ε, Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εργαστεί για πολλά χρόνια ως δημοσιογράφος για ελληνικές εφημερίδες όπως η Αυγή, το Βήμα. για τον ε, ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα, για το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ως, αντι... Ε, ανταποκρίτρια και επίσης για διάφορες άλλες εφημερίδες το 2000 2000 πήρε το ελληνοτουρκικό βραβείο δημοσιογραφίας για την ε, συμβολή της στην προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών. Και απονεμήθηκε το βραβείο αυτό στην Άγκυρα το 2000 από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, τον Αγέριο Παπανδρέο και τον Ισμαήλ Τζέμ. Η κυρία Ποδηματά είναι δημοσιογράφος, παραμένει δημοσιογράφος και με μεγάλη χαρά θα ανταλλάξει απόψεις μαζί σας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γενικότερα και η Ευρώπη αντιμετωπίσουν και θα αντιμετωπίσουν μετά από τις εκλογές. Αν έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη για τα θερμά λόγια. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Πράγματι είμαι δημοσιογράφος. Κάποιος που έχει ξεκινήσει σαν δημοσιογράφος παραμένει πάντα δημοσιογράφος. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που είμαι μαζί σας. Πολύ λίγο καιρό, δύο εβδομάδες πριν από τις ε, τόσο κρίσιμες ευρωεκλογές της 22ης και την 25η Μαΐου του 2014 Πιστεύω ότι αυτές οι ευρωεκλογέ είναι ίσως οι πιο κέρδιες, οι πιο κομβικές ευρωεκλογέ που έχουν λάβει ποτέ χώρα από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί το θέμα το οποίο θέλω να σας αναπτύξω, αφού κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις καταρχήν, και θα είμαι στη συνδιαθεσή σας για να έχουμε ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων, το θέμα λοιπόν το οποίο θέλω να σας παρουσιάσω σχετίζεται με τις ε, προκλήσεις που θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από τις εκλογές. Να ξεκινήσω τονίζοντας ότι είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι ένα είναι το κύριο διακύβευμα, η κύρια πρόκληση θα έλεγα ότι είναι και μια ιστορική πρόκληση για τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το ευρωπαϊκό εγχείρημα ως σύνολο και πρόκειται για το πώς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα μπορέσουν να αποκριθούν στις ανησυχίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών και αυτό μπορεί να σας φαίνεται προφανές. Αλλά το επαναλαμβάνω, γιατί πιστεύω ότι συμμεριζόσαστε και εσείς την άποψη ότι τα τελευταία πέντε χρόνια και ίσως αναπόφευκτα η Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν τις αστοχίες και τις δυσκολίες που προκλήθηκαν στις αγορές για να εμποδίσουν την επέκταση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Έχουμε καταφέρει να σταθεροποιήσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Έχουμε αποφύγει τα χειρότερα σενάρια σε ό,τι αφορά την κρίση. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε υποστεί σημαντικές απώλειες αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια και πέρα από τις σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές αρνητικές συνέπειες υπάρχει μια περαιτέρω σημαντική απώλεια που έχει να κάνει με την προηγούμενη πρόκληση που ανέφερα έχει προκύψει μια έλλειψη εμπιστοσύνη. Τα τελευταία λοιπόν πέντε χρόνια εμείς πρέπει να, θεωρήσουμε, πρέπει να θεωρήσουμε ότι υπήρξε αυτή η απώλεια όσο εμείς εστιάζαμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της, των αγορών. Το πετύχαμε αυτό μεν, πιστεύω θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει πολύ περισσότερα, αλλά συγχρόνως η διαδικασία αυτή οδήγησε και σε μια απώλεια εμπιστοσύνης. Δεν είχαμε την απαραίτητη εμπειρία ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δεν είχαμε εδρεωμένους μηχανισμούς και πολιτικές στο οπλοστάσιο απαντήσεων που θα έπρεπε να δώσουμε σε αυτή την ανευπροηγουμένου κρίση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η, επομένη, η πιο σημαντική πρόκληση για τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς το ευρωπαϊκό εγχείρημα ως σύνολο. Πέραν λοιπόν των απολειών που είχαν να κάνουν με την εμπιστοσύνη των πολιτών, ξέρετε ότι το κύριο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, είναι το θέμα της ανεργίας. Έχουμε πάνω από 26 εκατομμύρια άτομα που είναι άνεργοι, 5 εκατομμύρια νέοι που είναι άνεργοι και επειδή έρχομαι από την Ελλάδα θέλω να τονίσω ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη, στη δική μου χώρα, στην Ισπανία, τα ποσοστά ανεργίας έχουν ξεπεράσει το 25% του ενεργού πληθυσμού. Σε ορισμένε περιπτώσει για τους νέους έχουν ξεπεράσει και το 50%. Πιστεύω λοιπόν ότι τα δύο αυτά θέματα, το θέμα της απώλειας εμπιστοσύνης και οι κοινωνικές και οικονομικές απώλειες, είναι αλληλένδετα. Τα οικονομικά αυτά και κοινωνικά προβλήματα έχουν τροφοδοτήσει ανησυχίες και σκεπτικισμό έναντι του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της, να ε, ανακτήσει ένα λόγο ύπαρξη, ένα raison d'être στα μάτια των πολιτών, γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ μια ενωμένη Ευρώπη, η οποία θα μπορέσει να εκπληρώσει τις προσδοκίες των πολιτών της, είναι κατά τη δική μου άποψη η μόνη απάντηση. Όχι μονάχα για να βγούμε από την οικονομική κρίση, αλλά και να αντιμετωπίσουμε την παγκοσμιοποίηση. Δεν υπάρχει λοιπόν εναλλακτική λύση για μια από μια ενιαία Ευρώπη που μπορεί να δώσει απάντηση σε όλες αυτές τις ανησυχίες και τα ερωτήματα και πρέπει φυσικά να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι αναδύονται όλο και πιο πολλές αντιευρωπαϊκές ε, πολιτικές τάσεις, αυξάνεται ο εξτρεμισμός στις, αγορές, στις ε, κοινωνίες μας συγγνώμη, και επομένως η σημαντικότερη πρόκληση και το διακύβευμα των επόμενων πέντε χρόνων είναι το κατά πόσο θα εξασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία και οι ευρωπαίοι πολίτες θα δώσουν εντολή για περισσότερη και όχι για λιγότερη Ευρώπη. Και όπως ξέρετε η απάντηση αυτή θα δοθεί σε λίγες μέρες με τις ευρωεκλογές από τους πολίτες της Ευρώπης οι οποίοι συγχρόνως θα αποφασίσουν και για την ποσότητα και την ποιότητα των ε, δυνάμεων των πολιτικών που θα είναι υπέρμαχες της Ευρώπης ή αντίμαχες της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σίγουρα παρακολουθείτε τις δημοσκοπήσεις, αν λάβουμε υπόψη τις δημοσκοπήσεις σε σχέση με τις επικείμενες εκλογές, γνωρίζετε ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών θα υποστηρίξουν φιλοευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, φιλοευρωπαϊκές λύσεις, Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι γνωρίζετε ότι το ποσοστό των εξτρεμιστικών κομμάτων που αντικατοπτρίζονται στον αριθμό των μη εγγεγραμμένων στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, αυξάνει η δύναμη αυτών λοιπόν των πολιτικών δυνάμεων και αυτό δείχνει ότι αναδύεται, ότι αυξάνεται ο ευρωσκεπτικισμός που είναι ουσιαστικά ένα αμάλγαμα αντιευρωπαϊσμού και εξτρεμισμού στο πολιτικό στερέωμα. Με τα στοιχεία λοιπόν του Ευρωβαρόμετρου, με τις τελευταίες <clears throat> δημοσκοπήσεις που προέκυψαν από το Ευρωβαρόμετρο, μπορούμε να πούμε ότι χωρίς αμφιβολία βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ιστορικό παράδοξο. Ένα μεγάλο ποσοστό, μια πλειοψηφία των πολιτών μας πάνω από 70% από τη μία πλευρά δηλώνουν ότι αυτά που μας κρατούν ενωμένους στην Ευρώπη είναι πιο σημαντικά και περισσότερα από αυτά τα οποία μας χωρίζουν και επίσης μια μεγάλη πλειοψηφία πάνω από 50% λένε ότι μια ενιαία ενωμένη Ευρώπη μπορεί να προστατέψει και να δώσει περισσότερα ωφέλη στις ευρωπαϊκές κοινωνίες σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, παρά τα ενδιαφέροντα και ενθαρρυντικά αυτά στοιχεία, βλέπουμε ότι τα άκρα έχουν ενισχυθεί. Ενώ λοιπόν οι πολίτες μας θέλουν περισσότερη Ευρώπη, συγχρόνως, βάσει της δικής μου τουλάχιστον ερμηνείας, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας εκφράζει την απογοήτευσή του για τις αποτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζει πολιτικές δυνάμεις οι οποίες στην πραγματικότητα θέλουν να αποδομήσουν το συνολικό ευρωπαϊκό εγχείρημα και να το θέσουν ένα αμφιβόλο. <clears throat> Αν επιβεβαιωθούν λοιπόν αυτές οι τάσεις οι οποίες διαγράφονται από τις δημοσκοπήσεις, τότε θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου η λήψη απόφασης η λήψη αποφάσεων και όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο συνολικός μηχανισμός λήψης απόφασης θα επηρεαστεί και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη περισσότερο στο μέλλον ο ρόλος και οι θέση των αντιευρωπαϊκών δυνάμεων. Αυτό είναι λοιπόν το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και η Κομισιόν. Η νέα λοιπόν Κομισιόν η οποία θα προκύψει από τις ε, εκλογές, ξέρετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει πολύ πιο έντονο ρόλο στην διαμόρφωση της ε, Κομισιόν μέσω της εκλογής του Πρόεδρου της Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Συμβούλιο με τον νέο Πρόεδρό του θα πρέπει να λειτουργήσει σε αυτό το νέο πλαίσιο και να αντιμετωπίσει τα ανοιχτά μετώπα που υπάρχουν ενώπιόν μας. Κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα μετώπων που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα στην επόμενη θητεία της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την επόμενη πενταετία, απόλυτη προτεραιότητα για μένα είναι τα θεσμικά ζητήματα όπως η βελτίωση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας κάτι το οποίο για μένα σημαίνει μεγαλύτερη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, μεγαλύτερη συμμετοχή και μεγαλύτερη λογοδοσία. Για όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό σημαίνει ένα πιο στεναρό και ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερον, γνωρίζετε ότι λόγω των αποτυχιών στον οικονομικό στίβο, λόγω της έλλειψης καταλήλων μηχανισμών και πολιτικών για να αντιμετωπιστεί αυτή η τόσο σοβαρή οικονομική κρίση. Έχουμε αλλάξει και έχουμε πιστεύω βελτιώσει το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η πρόκληση για την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου είναι να εξασφαλίσουμε όχι μόνο θα λειτουργήσει το νέο αυτό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά ότι θα λειτουργήσει και συγχρόνως θα λειτουργήσει με μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία. Και με τον τρόπο αυτό και πάλι θα πρέπει να εξασφαλιστεί με μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και με μεγαλύτερη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διαδικασία αυτή. Αυτό λοιπόν είναι το θεσμικό τμήμα των προκλήσεων που βρίσκονται ενώπιόν μας για την επόμενη πενταετία. Υπάρχουν όμως παράλληλα και σημαντικές προκλήσεις σε σχέση με το μείγμα πολιτικών που πρέπει να ακολουθηθεί στο μέλλον, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια χωρίς προηγούμενο και μια απαράδεκτη ανεργία, ένα απαράδεκτο επίπεδο ανεργία, ιδίω σε ό,τι αφορά του νέου. Και εδώ πιστεύω ότι η κύρια, η κέρια πρόκληση για τα επόμενα χρόνια είναι να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης. Πρέπει με κάθε τρόπο να αποφύγουμε αυτό το οποίο λέγεται jobless recovery, δηλαδή μια οικονομική ανάκαμψη χωρίς όμως δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, βασιστούμε στα πρώτα ψήγματα ανάκαμψης που είναι ακόμα εύθραυστη που παρατηρούμε σήμερα και να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει βιώσιμη αυτή η ανάκαμψη και κυρίως με κύρια προτεραιότητα τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Η Ευρώπη, όπως ξέρετε, είναι το μόνο τμήμα του κόσμου όπου η οικονομική ανάκαμψη δεν έχει επανέλθει μετά από την ε, παγκόσμια οικονομική κρίση. Γι' αυτό σας λέω ότι βρισκόμαστε σε ένα δρόμο ανάκαμψης ο οποίος είναι ακόμα πολύ εύθωστος. Ξέρετε ότι διάφορες πολιτικές παρατάξεις, διάφορες πολιτικές οικογένειες έχουν διατυπώσει διαφορετικές προτάσεις για τα θέματα αυτά. Αυτό όμως το οποίο θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα είναι ότι πέραν αυτών των διαφορετικών προτάσεων υπάρχουν σημαντικές διαφορετικές, αντιμε... αντιμετωπίσεις μεταξύ αυτών που θέλουν πιο εθνικές προσεγγίσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα τα οποία σας προανέφερα και ακριβώς υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θέλουν περισσότερες λύσεις ευρωπαϊκές, περισσότερες απαντήσεις ευρωπαϊκές. Οπότε έχουμε ε, αυτού του είδους την ε, διχογνωμία ε, της αντίληψης των πραγματών γιατί από μια μεριά έχουμε εκείνους που πιστεύουν ότι η διέξοδος από ε, σημερινή κατάσταση είναι η επανεθνικοποίηση των πολιτικών και από την άλλη μεριά είναι τα κόμματα τα φιλοευρωπαϊκά, οι δυνάμεις φιλοευρωπαϊκές ε, που παρά τις ε, κατά τα άλλα διαφορετικές ιδεολογικές τους διαφορές θεωρούν ότι η λύση έγκυται στην Ευρώπη στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τελευταίο τώρα το οποίο θα ήθελα να σας αναφέρω Ήδη θα έρθει η Επίτροπος ε, Χιλντεγκάρ που είναι η υπεύθυνη για την κλιματική αλλαγή και θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω και να τονίσω το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την προηγουμένη κοινοβουλευτική θητεία έλαβε λοιπόν ρόλο πρωτοπόρο για την αντιμετώπιση το προβλήματων της αλλαγής του κλίματος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαμορφώσει την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το τόσο κρίσιμο ζήτημα του εγγύς μέλλοντος. Και εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε να συνεχίσει η Ευρώπη να είναι πρωτοπόρα στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος που είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σημαντικό το οποίο σχετίζεται φυσικά με την ενεργειακή πολιτική με την εξασφάλιση της προμήθειας της ενέργειας, την ε, αυτάρκεια σε σχέση με την εισαγωγή ενέργειας και επίσης το τελευταίο ε, το οποίο έχει να κάνει με την κρίση στην Ουκρανία η οποία όλο ένα και παροξύνεται και επιδεινώνεται που πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα, ακόμα ένα ενισχυτικό μήνυμα του γιατί η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει και να έχει και για τις ιστορικές υποθέσεις μια κοινή και ισχυρή φωνή. Τα σχετικά με τους μετανάστες επίσης κατέδειξαν ότι χρειάζεται κοινή πολιτική για την μετανάστευση ούτως ώστε να κατοχυρωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων αλλά επίσης και να είναι δίκαιη η κατανομή των αρμοδιοτήτων και βαρών μεταξύ των κρατών μελών. Οπότε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει πιστικές απαντήσεις για όλα αυτά τα αμέσως επόμενα χρόνια. Εάν θέλουμε να μπορέσουμε να επηρεάζουμε το παγκόσμιο γίγνεσθε και να μην θέλουμε να δούμε το ρόλο μας συρρυκνωμένο. Αλλά τέλος πάντων για να επιστρέψω στην αρχή των ε, όσων σας ανέφερα θα πρέπει να δώσουμε πιστικές απαντήσεις. Και για όλα αυτά τα προβλήματα νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει τη δρομή μας πολύ πιο νωρίς και όχι μετά τις εκλογές για να μπορέσουμε τη σημαντικότερη πρόκληση να αντιμετωπίσουμε αυτή που είπα στην αρχή. Δηλαδή την πρόκληση του να μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη, ε, την καρδιά των πολιτών, την εμπιστοσύνη προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, προς το σύνολο του ευρωπαϊκού οράματος. Αυτά, Γιάννη, και βεβαίως ε, πρόθυμα να απαντήσω τις τυχόν ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Νομίζω πως μετά από αυτή την εισαγωγή θα έχετε ερωτήσεις. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια σύνοψη, το βασικό δίλημα είναι μεταξύ αυτών που είναι υπέρ περισσότερων εθνικών λύσεων και όσων είναι υπέρ μιας πιο ευρωπαϊκής προσέγγισης. Πριν σας δώσω τον λόγο, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως έχουμε διερμηνία στα γερμανικά, ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, ολλανδικά, πολωνικά και ρουμανικά. Οπότε, έχετε τον λόγο. Ε, πριν κάνετε την ερώτησή σας, παρακαλώ να αναφέρετε το όνομα και το, το όνομά σας και το μήνυμα στο οποίο εργάζεστε. Ποιος θα ξεκινήσει. Παρακαλώ. I'm not sure. Oh, ναι, ωραία. Κύριε από την Γερμανία επισημάνατε πως ε, είναι σημαντικό να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Υπάρχει κάποια σχετική στρατηγική για το πώς θα γίνει αυτό. <coughs> Well, since uh, Κοιτάξτε, μιας ε, που γίνεται αυτή η συζήτηση 15 μέρες ε, πριν τις ε, ευρωεκλογέ. εγώ δεν το ανέφερα γιατί νόμιζα το είχαμε πει και νωρίτερα αλλά πάνω απ' όλα το κύριο μήνυμα πρέπει να είναι πως επαφίεται στους πολίτες να αποφασίσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εκλογές το εάν θέλουν ισχυρότερη Ευρώπη ή όχι και βεβαίως τι είδους Ευρώπη θέλουν τι πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξει στην Ευρώπη γιατί εγώ επέμενα πως η απάντηση κατά την άποψή μου όσον αφορά την βιώσιμη ε, διέξοδο από την κρίση τι εννοώ με αυτό δηλαδή μια διέξοδος η οποία θα μείωνε τις ε, πιθανότητες ανάλογης κρίσης στο μέλλον και αυτό σημαίνει να αντιμετωπίσουμε τους λόγους που μας οδήγησαν στην κρίση και βεβαίως σημαίνει επίσης πως ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά προτεραιότητα τώρα που αποφύγαμε τα χειρότερα με τις ε, απώλειες ε, που ανέφερα να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές και κοινωνικές ε, απώλειες που συνδέονται κατά την αποψή μου με, την, με το ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται πλέον την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει να μειωθεί η ανεργία, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Να Ευχαριστούμε για μια ανάκαμψη που θα τους περιλαμβάνει όλους που θα μειώσει τις ε, μακροοικονομικές ανισορροπίες π.χ. μιλάω τώρα για την Ευρωζώνη που ήταν ένας από τους λόγους ε, της κρίσης Αυτές ήταν κάποιες από τις ελλείψεις ε, στη λειτουργία της ΟΝΕ τα τελευταία δέκα χρόνια πρέπει λοιπόν νομίζω να δώσουμε λύσεις και απαντήσεις που θα πείσουν τους πολίτες ότι η ευρωπαϊκή οικοδόμηση είναι η μόνη απάντηση που μπορεί να δώσει τις αναγκαίες ε, λύσεις για το αύριο για στις, ε, στην καθημερινή ζωή για τις σημερινές και τις ευρεανές γενιές και νομίζω πως Αυτό παρά τις ε, δυσκολίες ε, της τρέχουσας ε, περίοδου είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξηγηθεί και εσείς, εμείς και εγώ βεβαίω. συμπεριλαμβάνω και εμένα στους δημοσιογράφους πρέπει να εξηγήσουμε το γιατί μια Ενωμένη Ευρώπη που έχει να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις ε, αυτές είναι το μόνο πλαίσιο που μπορεί να δώσει στους πολίτες στο βορρά, στον νότο, στην Ανατολή και στη δύση της Ευρώπης ένα πλαίσιο για να αντιμετωπίσουν τις ε, προκλήσεις ε, του σημερινού παγκοσμιοποιημένου κόσμου και των παγκοσμιοποιημένων προβλημάτων. Όχι μόνο στο επίπεδο των ε, χρηματαγορών, αλλά και στο επίπεδο του περιβάλλοντος ε, της κλιματικής αλλαγής. Νομίζω πως οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προωθήσουμε τα, τελευταία, τα επόμενα πέντε χρόνια πρέπει να υπάρξει μια τροποποίηση των πολιτικών ε, για τις οποίες είναι αναγκαία η Ευρώπη. Π.χ. η Ευρώπη πρέπει να εμπλακεί πολύ περισσότερο στα μεγάλα ζητήματα πολιτικής. Γι' αυτό ανέφερα την ανεργία, την κλιματική αλλαγή, την ε, ανάκαμψη που να τους περιλαμβάνει όλους ε, και όχι τόσο πολύ το να παρεμβαίνει σε, επίπεδα που πιο σε ζητήματα που πιο αποτελεσματικά αντιμετωπίζονται σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτούμε, να αποφασίσουμε το ότι χρειαζόμαστε πιο ισχυρή Ευρώπη, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει η Ευρώπη να μπλέκεται στα πάντα. Πρέπει να δούμε την κατανομή πολιτικών εκεί δηλαδή που χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και που χρειαζόμαστε ίσως λιγότερη Ευρώπη. Σε ευχαριστούμε Άννη. Επόμενη ερώτηση. Ναι, Κυριακή. Πατρίσια Βιέγερα από την Πορτογαλία. Λέτε πως οι εκλογές αυτές είναι διαφορετικές ε, λόγω του θέματος με τον πρόεδρο της Κομισιόν αλλά μήπως είναι διαφορετικές ε, γιατί είναι και ένα δημοψήφισμα για το ευρώ και την οικονομική πολιτική που έχει ακολουθηθεί και στη, για την πολιτική της Τρόικας που έχει επιβληθεί σε κάποιες χώρες. Ευχαριστώ. Ναι. Νομίζω πως ε, αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά όχι μόνο λόγω του ότι το Κοινοβούλιο θα μπορεί να επηρεάσει άμεσα την εκλογή του Πρόεδρου της Επιτροπής αλλά και λόγω των συνθήκων της περιραίουσας ατμόσφαιρας. Γι' αυτό επέμεινα στο ότι η βασική πρόκληση εδώ πέρα είναι να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Δημοψήφισμα τώρα εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη δημοψήφισμα. Γιατί ε, εντάξει αντιλαμβάνομαι και εγώ από την Ελλάδα είμαι εσείς από την Πορτογαλία. Και έχω δει πραγματικά την απογοήτευση, την οργή μεγάλων ε, κομμάτων, κομματιών με συγχωρείτε, κοινωνίας για τις επιπτώσεις της κρίσης. Από την άλλη θεωρώ πως δεν θα πρέπει να κάνουμε επιλογές ε, βασιζόμενοι στο θυμικό. Γιατί? Γιατί θεωρώ πως υπάρχει κίνδυνος εάν ε, το κίνητρο είναι όπως είπα συναισθηματικό να κάνουμε λανθασμένες επιλογές. Οπότε το βασικό εδώ πέρα δεν είναι να τιμωρήσουμε την Ευρώπη επειδή θεωρούμε σωστά ή όχι ότι η Ευρώπη μας τιμώρησε. Το σωστό νομίζω και η κρίσιμη απάντηση είναι το τι χρειάζεται να αλλάξουμε στην Ευρώπη για να δοθούν καλύτερες λύσεις από την Ευρώπη στα προβλήματα μας. Γι' αυτό εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη δημοψήφισμα. Γιατί αυτό το οποίο έχουμε σήμερα ως ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ως διαδικασία λήψης αποφάσεων, ως μείγμα πολιτικής ε, είναι το ιδεώδες. Όχι. Όπως είπε και ο Γιάννης, εγώ ανήκω σε μια πολιτική οικογένεια, έχω συγκεκριμένες ε, απόψεις ε, όσον αφορά το τι πρέπει να αλλάξει στην Ευρώπη. Από την άλλη, θεωρώ πως είναι επικίνδυνο να ευθύσουμε μια προσέγγιση του στυλ ναι ή όχι στην Ευρώπη. Κατά την άποψή μου η Ευρώπη είναι η απάντηση. Η Ευρώπη μας βοήθησε να αποφύγουμε τα χειρότερα και μιλάω και ως Ελληνίδα πολίτης παρά τις τεράστιες ε, ζήμιες ε, στην ε, οικονομία και στην κοινωνία για τις οποίες υπάρχουν και εθνικές και ευρωπαϊκές ευθύνες, όχι μόνο στη διαχείριση της κρίσης, αλλά και στο πώς ε, λειτουργούσαμε και πριν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πώς ε, οικοδομήθηκε η ΟΝΕ. Όλα αυτά ε, είναι, διαφορε... είναι διάφορες ελλείψεις και αποτυχίες. Και το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις σημαίνει πως έχουμε ευθύνη όλοι ειδικά όσοι διαμορφώνουν α, την πολιτική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να προσπαθήσουν να δώσουν τις σωστές απαντήσεις ε, για να αντιμετωπίσουν ακριβώς αυτές τις ελλείψεις. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες να αποφασίσουν ε, λογικά με το μυαλό το τι, με τη λογική το τι είδους ε, Ευρώπη θέλουν να κάνουν ε, τις ανάλογες επιλογές σε εκλογές. Ευχαριστώ Άννη. Επόμενη ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Αντρέη Μασέκα από την Σλοβακία. Σε ποιους τομείς χρειαζόμαστε περισσότεροι και σε ποιους τομείς λιγότερη Ευρώπη, όπως είπατε. Μπορείτε να μας πείτε κάποια σημεία στα οποία χρειαζόμαστε λιγότερη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Yes, um, ναι. Πού χρειαζόμαστε πιο πολύ Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανείς. Πιστεύω ότι πρέπει να προωθήσουμε μια γνήσια Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως θα έλεγα. Μέχρι στιγμής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εργαστεί περισσότερο στο νομισματικό πυλώνα. Είχαμε ένα κοινό νόμισμα που ήταν ένα είδος ορφανού νομίσματος γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα κυριαρχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε δημοσιονομικά παραδείγματο χάρη θέματα, γιατί αυτή παρέμενε στο εθνικό επίπεδο. Είχαμε μια κεντρική τράπεζα με πολύ περιορισμένες εξουσίε, με περιορισμένη εντολή. Και έχουμε πετύχει κάποια πρόοδο στα θέματα αυτά. Γι' αυτό αναφέρομαι στο νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το οποίο εισήχθη πρόσφατα και παίζει σημαντικό ρόλο τη δημιουργεί διαδικασίες για τη δημοσιονομική διαδικασία συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δίδει και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για καλύτερο οικονομικό συντονισμό. Ένα άλλο παράδειγμα θα προτιμούσα ορισμένα θέματα τα οποία είναι ταμπού προς το παρόν. Τα θέματα φορολογίας, του χάρη, θα πρέπει να τεθούν σε συζήτηση. Και να, θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση στα θέματα αυτά. Και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο η διαδικασία λήψης απόφασης σε αυτό το τομέα τον πάρα πολύ ευαίσθητο είναι η σωστή. Πιστεύω ότι θα πρέπει ότι θα πρέπει να τροποποιήσουμε τον κανόνα της ε, ομοφωνίας γιατί στον τομέα αυτό στην πράξη δεν αφήνει η, η ανάγκη ομοφωνίας να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες μπορούν να κινούνται προς το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Θεωρώ λοιπόν ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την Τραπεζική Ένωση είναι πραγματικά ιστορικού χαρακτήρα. Έχουν παίξει σημαντικό ρόλο η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν είχε μια ευρεία συνένεση στα θέματα αυτά με όλες τις πολιτικές ομάδες να έχουν επιφυλάξεις για την τελική συμφωνία που ελήφθη για την Τραπεζική Ένωση. Επομένως αυτό το οποίο θέλαν ήταν να είναι πιο φιλόδοξη η απόφαση αυτή για την Τραπεζική Ένωση. Φυσικά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι είναι μια ιστορική απόφαση η οποία έχει και τη δυνατότητα κατά τη δική μου άποψη να αντιμετωπίσει πολλές ε, δυσλειτουργίες που είχαμε στο παρελθόν σε ό,τι αφορά της χάρη το να ξεπεράσουμε την, ε, τον κατακαιρματισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα και του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη που είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα κύρια εμπόδια στο δρόμο για μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση. Αυτές λοιπόν είναι περιπτώσεις και παραδείγματα όπου τονίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε προς μια πιο ισχυρή Ευρώπη και παράλληλα να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους αυτή η Ευρώπη θα είναι πιο δημοκρατική και πιο υπόλογη στους πολίτες της. Είναι πολύ σημαντικά λοιπόν αυτά να τα προσπαθήσουμε να τα επιτύχουμε, να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις που αυξάνουν την ε, λογοδοσία και την ε, διαφάνεια στη διαδικασία λήψης απόφασης. Ναι, δεν έχω εύκολες απαντήσεις σε όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχουν όμως πολλά πράγματα που πιστεύω ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο εποφελώς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχουν θέματα όπου οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι πολύ πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των κοινωνιών μας. Και η διαδικασία λήψης απόφασης σε όλα αυτά τα θέματα που έχουν ε, τοπική, τοπικό χαρακτήρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με μία συνολική διαδικασία Πολλέ φορέ αντιμετωπίζοντα με, με ένα μονοκόμματο τρόπο τα προβλήματα, δημιουργούμε σοβαρότερα προβλήματα. Ευχαριστώ, Άννη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Γκρέγκορ Ντεκλέρ, είμαι μεγάλο δημοσιογράφο στην Ματά, ε, στην εφημερίδα Ματά. <clears throat> Δύο ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, σε, απευθύνομαι σε εσά ω ε, πολίτη της Ελλάδος. Θυμάμαι την εποχή που η Νικόλ Φοντέν ήταν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν εισήχθη το ευρώ και είπε το να μπει η, η Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Τι πιστεύετε γι' αυτό. Δεύτερον, φαίνεται ότι οι πολίτες περιμένουν από την Ευρώπη στο κοινωνικό επίπεδο πολλά. Μπορείτε να φανταστείτε ένα ελάχιστο μισθό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το αντίστοιχο του γαλλικού ΣΜΙΚ. Μπορείτε να επαναλάβετε το δεύτερο τελευταίο τμήμα της να καθιερωθεί, να θεσπιστεί ε, ελάχιστος μισθός, ελάχιστο μερομίσθιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Α, σμικ, σμικ. Α, σμικ. Bon. Est-ce que euh, c'était une erreur pas de... Δεν ξέρω αν ήταν λάθος ή όχι το να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα. Επάνω σε αυτό Έχω δύο να σας πρώτα. Πρώτα δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει σε όλη την περίοδο που μας έχει χτυπήσει η κρίση γιατί αυτό το οποίο εγώ το ονομάζω ότι είναι μια ολόκληρη πολεμική ε, δηλαδή το να κατηγορούμε να κουνάμε το δάχτυλο και να βάζουμε τον έναν απέναντι στον άλλο ε, αυτό ήταν τελείως ε, αντιπαραγωγικό σε αυτή την περίοδο της κρίσης. Και αντίθετα θεωρώ ότι τέτοια σχόλια και τέτοιες τοποθετήσεις αν ήταν δηλαδή λάθος να, να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα ε, ή ότι καλύτερα να διευκολύνουμε την έξοδο της ε, Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που αποκαλούμε εγκρέξιτ. Ε, όλα αυτά, όλα αυτά, κατά την απόψή μου, έχουν χειροτερεύσει την κατάσταση κατά πολύ και έχουν περιπλέξει την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης και έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Οπότε δεν θα σας το σχολιάσω, δεν θα σας απαντήσω σε αυτό, δηλαδή αν ήταν λάθος ή όχι. Όμως, θα ήθελα να επενθυμίσω το εξής. η απόφαση του να δημιουργήσουμε την οικονομική και νομισματική ένωση ήταν μία απόφαση που ελήφθη στα δεκαετία του 90 και αυτή η απόφαση ελήφθη όχι μόνο για οικονομικούς λόγους και με οικονομικά κριτήρια. Βεβαίως και όταν κανείς δημιουργεί μια τέτοια νομισματική ένωση επιβάλλεται να θεσπίζει και κάποιους ε, δημοσιονομικούς κοινού κανόνες. Αλλά ταυτόχρονα η απόφαση του να προχωρήσουμε προς την ημερία της ΟΝΕ ήταν απόφαση στρατηγική για την ε, Ευρώπη. Μια απόφαση που συνδέεται με το πώς τότε βλέπαμε τα πράγματα για τη διδικασία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Για το ποια πορεία θα πάρει η ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Η δημιουργία της ΟΝΕ ακριβώς όπως και η κρίση που αντιμετωπίζουμε την τελευταία πενταετία. Ιωνέ, ναι, λέγω. Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Έγινε αναπόφευκτα με τρόπο που δεν ε, οδήγησε στην ε, ολοκλήρωση της κατά 100% Ίσως ε, θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη τις βασικές μας εμπειρίες πάνω σε αυτό, αλλά η βασική προσέγγιση ήταν το να δημιουργήσουμε, το να θεσπίσουμε, να υιοθετήσουμε το κοινό ενιαίο νόμισμα το οποίο θα ήταν η ατμομηχανή για την οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πράγματα όμως δεν πήγαν πάρα πολύ καλά γιατί δεν προβλέψαμε 100% όπως έχω επισημάνει και όπως όλοι γνωρίζουμε το τι θα γίνει. Αλλά σας τα λέω αυτά γιατί κατά τη γνώμη μου ακριβώς τώρα αυτή την προτεραιότητα θα πρέπει να έχουμε. Να κάτσουμε και να σκεφτούμε τότε πάνω σε ποια βάση λάβαμε αυτή την ε, απόφαση που να έχουμε το κοινό νόμισμα. Οπότε να ξαναποκτήσουμε ως προτεραιότητα την στρατηγική διάσταση εκείνης της αποφάσεως. Και τώρα να αποπειραθούμε το να δώσουμε τις δέουσες απαντήσεις εκεί. τις απαντήσεις που δεν έχουμε μπορέσει να δώσουμε κατά την τελευταία δεκαετία. Εν πάση Για να αν... αναχθούμε στο γενικότερο ζήτημα του αν χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και ε, τι θα πρέπει να δώσουμε ως απάντηση στους Ευρωπαίους τώρα ενώπιση των εκλογών. Έχω να σας πω ότι για μένα είναι φανερό. Μια προβληματική που θα οδηγούσε στην συρρήκνωση του ρόλου της ΟΝΕ θα ήταν κάτι το καταστροφικό, κάτι το όλος διόλου λάθος. Μας οδηγούσε σε λάθος κατεύθυνση σε σχέση με τα συμπράσματα του οποία θα έπρεπε να έχουμε εξαγάγει κατά την ε, περίοδο της κρίσης. Οι απαντήσεις και οι λύσεις. Πού έγινε. Όχι στο να γίνουμε λιγότεροι το αντίθετο. Νομίζω θα πρέπει να πάρουμε κάποια μαθήματα, να εξαγούμε κάποια συμπεράσματα και έτσι να μπορέσουμε πιο αποτελεσματικά να εκμεταλλευτούμε τις ε, δυνατότητες που έχουν ε, τα κράτη-μέλη, όσοι συμμετέχουν στην ΟΝΕ, ε, όσοι συμμετέχουν γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ελάχιστο εισόδημα, το ελάχιστο μισθό. Ε, εγώ είμαι σοσιαλδημοκράτης και βεβαίως είμαι 100% υπέρ μιας τέτοιας πρότασης, κάτι το οποίο άλλωστε ε, περιέχεται ε, στο προεκλογικό μας πρόγραμμα για τους ευρωπαϊκούς τους σοσιαλδημοκράτες, το να θεσπιστεί ελάχιστος μισθός σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Γενικότερα, επιμένουμε, τονίζουμε την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης, ούτως ώστε να καλύψουμε και τα κοινωνικά ζητήματα σε αυτή τη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου. έτσι να δημιουργηθεί αυτός ο οικονομικός και κοινωνικός πυλώνας. Η επόμενη ερώτηση. Ναι, από εδώ μια ερώτηση. Καλημέρα. Μίχο, Ρωμάνος για την Ρωμανία Λίμπερα. Για πες μας κάτι για το μέλλον. Εάν οι αντιευρωπαϊστές, εάν οι ακροδεξιοί, αυτά τα κόμματα τα καταφέρουν και πάνε καλά στις ευρωπαϊκές εκλογές. Θα συγκροτήσουν μια καινούργια πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσείς θεωρείτε ότι ελοχεύει ο κίνδυνος οι παραδοσιακές πολιτικές οι οι σοσιαλιστές, το Λαϊκό Κόμμα ε, να συρρυκνωθούν στο μέλλον και να ενδιαφέρονται λιγότερο στο να παλεύουν για το ευρωπαϊκό όραμα για να θέλουν ε, ε, περισσότερη Ευρώπη. Γιατί τότε θα χρειάζεται να αλλιεύσουν ψήφους. Σας ευχαριστώ. Όχι, όχι, εγώ θεωρώ ότι οι μεγάλες πολιτικές ε, φιλοευρωπαϊκές οικογένειες και κυρίως βεβαίως μιλώ για τη δική μου πολιτική οικογένεια, αλλά δεν ισχυρίζομαι ότι αποκλειστικά εμείς είμαστε οι συνήγοροι, οι υπερασπιστές του Ευρωπαϊκού Οράματος, οπότε ε, το γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και ότι είναι ενισχυτική η αύξηση της επιρροής των ε, ε, ακραίων αντιευρωπαϊκών δυνάμεων που έχει οδηγήσει σε περισσότερη αποφασιστικότητα από πλευρά αυτών των πολιτικών κοινωνιών. Σίγουρα πάντως αυτό ισχύει για τους σοσιαλδημοκράτες. Ούτως ώστε να προστατεύσουμε αυτό το οποίο δημιουργήσαμε αυτές τις δεκαετίες. Αυτό το υπέροχο ευρωπαϊκό όραμα που υπάρχει και θα πρέπει να εξηγήσουμε εκ νέου το πώς θα ήταν σήμερα ο κόσμος και η Ευρώπη αν δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί σας ξαναπαραπέμπω στα όσα γίνονται σήμερα στην Ουκρανία και καθίστε και σκεφτείτε και για το θέμα της ειρήνευσης και της ειρήνης γιατί υπάρχει μια πλειοψηφία πολιτών που θεωρούν ότι το θέμα, ο κίνδυνος πολέμου που ήταν ε, πηγή έμπνευσης ε, αιτία για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ε, θεωρούν επομένω ότι το πρόβλημα λύθηκε διαπαντός θεωρούν κάποιοι και ότι πια δεν κινδυνεύουμε να πέσουμε σε εμπόλεμη κατάσταση αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο και γι' αυτό και σας παραπέμπω στα όσα γίνονται στην Ουκρανία δεν θα πρέπει να διαπράξουμε το λάθος να πιστέψουμε ότι κάποια πράγματα είναι δεδομένα, αυτονόητα, γιατί γεννηθήκαμε υπό κάποιες τέτοιες ε, συγκεκριμένες περιστάσεις και συνθήκες. Γεννηθήκαμε σε περίοδο ειρήνης. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι δεν ελοχεύει ο κίνδυνος του πολέμου. Θα πρέπει επομένως αυτό να μην το ξεχνούμε. τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε η Ευρώπη, ποιο θα ήταν το κόστος της μη ύπαρξης της Ευρώπης. Σκεφτείτε, κυρίως σε επίπεδο ασφάλειας. Γι' αυτό και σας ανέφερα για τα γεγονότα της Ουκρανίας. Υπάρχουν και άλλα θέματα νομίζω ότι είναι πιο αποφασισμένες οι παραδοχές και πολιτικές οικογένειες γιατί ακριβώς αντιμετωπίζουμε αυτή την άνοδο της επιρροής αυτών που απορρίπτουν το ευρωπαϊκό όραμα την, την αύξηση του εξτρεμισμού και είμαστε 100% πεπισμένοι ότι τέτοιες προσεγγίσεις όπως εκείνες είναι καταστροφικές, είναι λαϊκιστικές. Δεν αρνούμε ότι ασκούν επίδραση εκείνες οι φωνές και οι δυνάμεις Ακριβώς ο λαϊκισμός σε περίοδο κρίσης έχει αποτελέσματα περισσότερο παρά σε μια φυσιολογική περίοδο. Όπως προανέφερα, είμαστε τώρα πολύ πιο αποφασισμένοι. Να δώσουμε τη μάχη και έτσι να προστατεύσουμε όχι μόνο ότι οικοδομήσαμε, αλλά και για να εξηγήσουμε ποια είναι η ωφέλεια, το κέρδος για την καθημερινή ζωή του κόσμου από αυτό το οποίο οικοδομήσαμε και να εξηγήσουμε ποιος θα ήταν ο κίνδυνος εάν η ευρωπαϊκή οικοδόμηση τεθεί ένα αμφιβόλο. Εάν επιλέξουμε να συρρυκνώσουμε, να ε, επιφέρουμε ε, υποβάθμιση της Ευρώπης στο μέλλον. Ευχαριστώ. άλλε δύο ερωτήσεις ε, θα ακούσουμε. Η κυρία έκανε ήδη μια ερώτηση. Οπότε, εσείς, ναι, από την Πορτογαλία, να έχετε ήδη κάνει ερώτηση. Να κάνει και κάποιο άλλο κάποια ερώτηση. Εσείς, λοιπόν, οι δύο. Και ο συνάδελφο εκεί στο βάθος. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα. Ιταλός δημοσιογράφος του είμαι. Υπάρχει ένα μανιφέστο κάποιων οικονομολόγων Γάλλων που λέει πως ε, το να έχουμε μία ενιαία δημοσιονομική πολιτική στην Ευρώπη θα είναι δυνατόν μόνο αν υπάρχει ένα ενιαίο κοινοβούλιο της Ευρωζώνης. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν την ε, άποψή σας. Αν μπορούμε δηλαδή να έχουμε κάποιο ενιαίο ευρωπαϊκό χρέος αντί εθνικό. Η δεύτερη ερώτηση. Βόλταν Λάιτσιχ ε, από την μεγαλύτερη εφημερίδα του Λουξεμβούργου, την Luxembourg Avot. Έχω μία ερώτηση ε, για το θέμα περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη και αναρωτιέμαι αν ε, ε, είχε γίνει στο παρελθόν σεβαστή επαρκώς η αρχή της επικουρικότητας. Καμιά φορά υπάρχει εντύπωση πως υπήρχε υπερβολική νομοθεσία για τα μικρά και ανεπαρκής νομοθεσία για τα μεγάλα. Ειδικά σε κάποιες ε, χώρες στην Ευρώπη που έχουν ανίσχυρες ή αναποτελεσματικές ε, κυβερνήσεις ε, περίμεναν από την Ευρώπη να περάσει νομοθεσία και να βελτιώσει τις οικονομικές και πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες ενώ σε άλλες χώρες όπου λειτουργεί σωστά το κράτος υπάρχει μάλλον η τάση να υπάρχει λιγότερη Ευρώπη ή να περιορίζεται η νομοθεσία στο απολύτως ε, απαραίτητο. Συμφωνείτε, παραδείγματος χάρη, πως στον τομέα της ανεργίας ε, ε, δεν επαφίεται στην Ευρώπη να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, αλλά πρέπει να δημιουργήσει τις συνθήκες, ένα σωστό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον για να μπορέσει να ανθίσει, να ανθίσουν οι επιχειρήσεις. Bon, donc euh, créer un parlement euh, euh, Για ένα κοινοβούλιο της Ευρωζώνης. Ναι, αυτό πραγματικά βρίσκεται στο επίκεντρο της προβληματικής ε, γενικότερα στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο κοινοβούλιο τελευταία διετία, τριετία, οπότε... Να είμαι ειλικρινής, πρέπει να σας πω ότι δεν έχω μια λύση για το πρόβλημα αυτό, η οποία να είναι μια εύκολη λύση, είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορέσαμε μέσα στην τρέχουσα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καταλήξουμε σε μια οριστική λύση παρά το γεγονό ότι έλαβαν χώρα πολύ έντονε και πλούσιε συζητήσει. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι σήμερα είμαστε 18 χώρε που είναι στη ζώνη του ευρώ και συμμετέχουν στην ε, Οικονομική αυτή και Νομισματική Ένωση. Σύμφωνα με τις συνθήκες όμως το ευρώ παραμένει το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η μεγάλη πλειοψηφία των άλλων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι στη ζώνη του ευρώ, εκτός από δύο χώρες οι οποίες έχουν προτιμήσει την αυτοεξαίρεση, το opt-out, όλες οι άλλες χώρες έχουν πάντα την προοπτική της εν καιρό προσχώρησης στην ζώνη του ευρώ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι τα πράγματα έχουν έτσι. Πιστεύω θα ήταν κάπως επικίνδυνο να δημιουργήσουμε θεσμούς οι οποίοι θα είχαν χαρακτήρα διαχωρισμού των διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατηγορίες. Από την άλλη πλευρά βέβαια το ενιαίο νόμισμα και η Οικονομική και Νομισματική Ένωση δημιουργούν de μία διάκριση μεταξύ των χωρών που είναι στη ζώνη του κοινού νομισματός και σε αυτών που δεν είναι, αλλά που δεν θα πρέπει να αποκλειστούν από, την, ε, από τον προβληματισμό για το ευρώ. Εγώ λοιπόν σας ε, τονίζω ότι μετά από πολλούς μήνες συζήτησης και αναλογισμού καταλήξαμε και φυσικά αυτό μπορεί να το αλλάξει το επερχόμενο κοινοβούλιο αποφασίσαμε να μην δημιουργήσουμε μια τέτοια δομή ένα κοινοβούλιο για τη ζώνη του ευρώ αλλά να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε, παραγωγικά χάρη με τη δημιουργία μιας υποεπιτροπής μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα αντιμετωπίζει τα θέματα της ζώνης του ευρώ, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και όπου θα συμμετέχουν όμως όλα τα μέλη χωρίς αποκλεισμό βουλευτών από χώρες που δεν είναι μέσα στην ε, ζώνη του ευρώ. Αλλά οι εισηγητές που θα εκθέσουν, που θα άπτονται της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης θα την χάνουν για αυτές τις ε, εισηγήσεις προτεραιότητα για την εκθέσει λοιπόν και για την προεδρία αυτής της υποεπιτροπής θα υπάρχει κάποια προτεραιότητα για τους βουλευτές οι οποίοι προέρχονται από χώρες της ζώνης του ευρώ. Δεν είναι ιδανική λύση βέβαια. Αλλά μπορεί να είναι και ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της καλύτερης λειτουργίας λύσεων που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα γιατί θα πρέπει να συνδυάσουμε την, τον μη αποκλεισμό των βουλευτών από τις χώρες που δεν είναι μέσα στη ζώνη του ευρώ με την άλλη επιτακτική ανάγκη να μπορούμε να έχουμε απαντήσεις σε τα ερωτήματα που αντιμετωπίζουμε με έναν τρόπο που θα είναι πραγματικά δημοκρατικός και να υπάρχει και ένα σύστημα λήψης αποφάσεων για τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να συνδυαστούν και με μια βελτίωση, μια κατεπηγόντως απαραίτητη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο γίνεται αυτή η λήψη απόφαση και κυρίως και με την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας για τις αποφάσεις του Eurogroup. Εδώ είναι ένας τομέας όπου πρέπει να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις. Και σε ό,τι αφορά την αρχή της επικουρικότητας. Δεν νομίζω ότι εξασφαλίζεται αυτή η αρχή σωστά έτσι όπως ε, αναφερθήκατε εσείς. Εγώ με την άποψή σας ότι παραδείγματο χάρη σε ορισμένου τομεί έχουμε πράγματι και απόλυτα δικαιολογημένα την εντύπωση ότι υπάρχει μια υπερβολική νομοθετική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λεπτομεριακά θέματα, ενώ συγχρόνως δεν υπάρχει αρκετή νομοθετική δραστηριότητα για θέματα τα οποία είναι πιο ουσιαστικά και όπου η Ευρώπη θα έπρεπε να παρεμβαίνει περισσότερο. Και αυτό ακριβώς προσπάθησα να σας περιγράψω στην αρχή της παρεμβασής μου, ότι χρειάζεται να σκεφτούμε ποια είναι η σωστή ισορροπία. Ποιες είναι οι αρχές οι οποίες πρέπει να πιτανεύουν πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν ποιε θα είναι οι πολιτικές οι οποίες κατά προτεραιότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα, γιατί η ευρωπαϊκή κλίμακα είναι πιο αποτελεσματική και ικανή να οδηγήσει σε καλύτερη αποτελέσματα, σε καλύτερα αποτελέσματα με τρόπο συνεκτικότερο και να μπορέσει με μεγαλύτερη ταχύτητα να καταλήξει σε λύσεις. Και από την άλλη πλευρά πια είναι τα θέματα και οι πολιτικές όπου οι τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές αρχές είναι σε καλύτερη θέση για να ρυθμίσουν τα θέματα αυτά και όπου πρέπει να ανακτήσουν κατά συνέπεια έδαφος. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα για την ε, επόμενη πενταετία μετά από τις ευρωεκλογέ. και αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της συνολικής συζήτησης για το τι είδους Ευρώπη θέλουμε να οικοδομήσουμε. Θέλουμε μια Ευρώπη η οποία θα δώσει απαντήσεις σε ποια προβλήματα. Ποια είναι η εικόνα μας λοιπόν, το όραμά μας για μια τέτοια Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να ανακατευθύνουμε την ε, πορεία μας. Θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η στάση μας εναντί της Ευρώπης στο μέλλον και ποιες θα πρέπει να είναι οι δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από τους νέους περιορισμούς οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί και πιστεύω ότι όλοι θέλουμε να έχουμε μια προσέγγιση και ένα όραμα το οποίο θα οδηγήσει στην ε, ανακατεύθυνση της ε, ευρωπαϊκής οικοδόμησης και δεν θα την εμποδίσει και έτσι θα μπορέσουμε να επανακαθορίσουμε την ισορροπία μεταξύ των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτών που είναι καλύτερα να αντιμετωπίζουν σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ, Άννη. Ας ελπίσουμε, πιστεύω ότι είναι πολύ καλό το συμπέρασμά σου, όταν μιλάς για νέους περιορισμούς, νέες υποχρεώσεις που δημιουργούνται για τη σχέση των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ότι έτσι πρέπει να ανα ναι, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μιας ε, δημοσιογράφου που είναι και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοσιογράφων που βρισκόνται στο κοινό. Σε ευχαριστώ, ήταν λύση η συζήτηση, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σας εύχομαι καλή συνέχεια. So, uh, a short announcement. So, Θα έχουμε και ένα έγγραφο το οποίο θα σας δοθεί για να απαντήσετε, για να δώσετε κάποια ανάδραση στα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν και περνάμε τώρα στο τρίτο τμήμα του σεμιναρίου, της πολιτικής πτυχίας της εκστρατείας.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 So, please, uh, take again Καθίστε, παρακαλώ. Και πάλι, μετά από το διαλυματάκι. Συνεχίζουμε με το τρίτο μέρος ε, του σεμιναρίου, ε, στο οποίο ο Ζαν Μεντούκο, πρόσωπος ε, του Κοινοβουλίου, και διευθυντής ΜΜΕ θα παρουσιάσει και θα συζητήσει μαζί σας τις πολιτικές πτυχές ε, της ε, εκστρατείας ε, και ταυτόχρονα θα σας παρουσιάσει τις τελευταίες τάσεις και προβολές της μελλοντική σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους. Θα είμαι σύντομος. Θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνοψη των ε, παρεμβάσεων τις οποίες ακούσατε. Τον Κλάους Βέλε, Χουαν Λαούς, ε, την ε, κυρία Ποδηματά, την Αντιπρόεδρο για να είναι τα πάντα σαφή. Μετά, 5-10 λεπτά στην τελευταία προβολή για τα πιθανά αποτελέσματα των εκλογών και μετά ευχαριστώ να απαντήσω στις ε, ερωτήσεις σας ε, κριτική απόψεις. Να σας πενθυμίσω κάποια νούμερα πρώτα απ' όλα για το τι έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία πέντε χρόνια. Όταν μας ρωτάει κανείς το γιατί είναι διαφορετικές αυτή τη φορά οι εκλογές. Ε, πάντα το πρώτο που λέμε είναι η εκλογή του Πρόεδρου της Κομισιόν, πράγματι, αλλά υπάρχουν και άλλα δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι πως ίσως λόγω της κρίσης, ίσως λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας, ίσως λόγω και των δύο αυτών στοιχείων η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ περισσότερες αρμοδιότητες και είναι πολύ πιο ορατή στους πολίτες από ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Αλλά υπάρχει άλλο ένα στοιχείο που επίσης είναι ενδιαφέρον, το ότι από τη Λισαβόνα και μετά το κοινοβούλιο έχει γίνει ένα πραγματικό κοινοβούλιο, ισχυρό και ε, με επιρροή. Όταν λέω με επιρροή, δεν μιλάω για απόψεις, ε, ψηφίσματα, η διαβούλευση με τους βουλευτές αλλά μιλάω για νομοθεσία κανόνες, οδηγίες ε, και τα λοιπά. Αυτό είναι νομίζω το πιο ενδιαφέρον σημείο από αυτή την άποψη το ότι δηλαδή την τελευταία πενταετία υιοθέτησε πάνω από 950 ε, πάνω από 950 νομοθετήματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγκρίνεται με οποιοδήποτε κοινοβούλιο στον κόσμο. Έχει εγκρίνει πάνω από 2.500 κείμενα, τροπολογίες δηλαδή και αλλαγές κειμένων, πάνω από 20.000 ε, ψηφοφορίες και πάνω από 1.500 ε, συναντήσεις στο πλαίσιο τριμερούς διαλόγου με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για να διαμορφωθεί η νομοθεσία πριν έρθει στο Κοινοβούλιο και στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου. Βέβαια αυτά είναι νούμερα, αλλά εάν δείτε την δεύτερη διαφάνεια και το ποιες ήταν οι βασικές στιγμές βλέπετε πως υπάρχει εδώ πέρα σοβαρή νομοθεσία δεν είναι τεχνικά ζητήματα έτσι ήταν η κατάσταση πριν από 20 χρόνια, δηλαδή το Κοινοβούλιο ψήφιζε αλλά πάντα για ε, κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Τώρα μιλάμε για πολιτική, για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 7 χρόνια, για τη μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής, ε, της πολιτικής αλληλείας, ε, των περιφερειακών ταμείων, για το ότι απορρίφθηκε η θέση ενισχύ τη συμφωνίας με τις Ηνωμένε Πολιτείε για την χρήση από τις ΙΠΑ όλων των δεδομένων από τραπεζικές συναλλαγές το ότι επίσης απέρριψε το Κοινοβούλιο την θέση ενισχύ της συνθήκης ΑΚΤΑ που ήταν κατά της ε, πειρατείας ε, και στο διαδίκτυο, η νομοθεσία περί περιαγωγής, ε, για τα στεγαστικά δάνεια, ευαίσθητο ζήτημα σε πολλές χώρες, για την Τραπεζική Ένωση και πολύ περισσότερο για την οικονομική ε, διακυβέρνηση. Τα διάσημα εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διπλά και εξαπλά πακέτα τα οποία επέτρεψαν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπληρώσει την νομισματική ένωση με μία αρχή οικονομικής ένωσης. Μετά, οι υποψήφοι είναι γνωστοί πλέον. Μία από τις ε, επιτυχίες, θα έλεγα, της εκστρατείας μέχρι στιγμής για τις ε, συζητήσεις ε, των υποψηφίων θα έχουμε και εδώ πέρα μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την οποία δεν οργανή το Κοινοβούλιο αλλά η EBU Eurovision στις 15 Μαΐου 9 το βράδυ και θα μεταδοθεί από τουλάχιστον 30 ευρωπαϊκά κανάλια και πολλά άλλα οπωσδήποτε που δεν είναι ευρωπαϊκά μου έκανε εντύπωση το ότι είδα παραδείγματος χάρη ότι θα μεταδοθεί στον Καναδά. και από χώρες που δεν είναι κράτη-μέλη. Αυτό είναι σημαντικό γιατί έτσι θα μπορέσουμε να δείξουμε στους πολίτες γιατί οι εκλογέ αυτές είναι διαφορετικές σε σχέση με το παρελθόν. Όσον αφορά τη νύχτα των εκλογών, ναι, θα είναι οπωσδήποτε μια μεγάλη υπόθεση για τα ΜΜΕ. Το 2009 υπήρχαν γύρω στους 500 δημοσιογράφους που παρακολουθούσαν τα αποτελέσματα ανά χώρα και βεβαίω ε, ήθελαν και μια γενικότερη ευρωπαϊκή εικόνα που την δίνει μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κανείς άλλος στην Ευρώπη δεν έχει την δυνατότητα να δώσει ε, το βράδυ των εκλογών την εικόνα αυτή. Αυτή τη φορά υπολογίζουμε πως θα έχουμε τον διπλάσιο αριθμό δημοσιογράφων γύρω στους χίλιους συναδέλφους σας, ίσως και κάποιοι από σας που θα δουλεύουν εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 25 και ίσως και στις 26 και στις 27 γιατί όπως είπε και ο κύριος Βέλε στις 27 θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συναντήσεις η μία εδώ στο Κοινοβούλιο η διάσκεψη των Προέδρων που σημαίνει ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου συν ή ε, επικεφαλής των πολιτικών ομάδων και το βράδυ η άτυπη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στις δύο περιπτώσεις για να δούμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το πώς θα οργανώσουμε τα επόμενα βήματα που συμπεριλαμβάνουν οπωσδήποτε και την ε, εκλογή του Πρόεδρου της Κομισιόν. Τώρα, να περάσω κάποιες διαφάνειες και θα φτάσω μέχρι σχεδόν την τελευταία που είναι μια προβολή. Αυτές είναι εβδομαδιαίες προβολές και αφορούν ε, τις καταρχήν τις έχουν προετοιμάσει οι υπηρεσίες μας εδώ με την βοήθεια της ε, TNS ε, μιας εταιρείας ε, δημοσκοπήσεων γαλλικής εταιρείας συνεργάζονται μαζί μας εδώ και 15 χρόνια είναι η τρίτη εκλογική αναμέτρηση που μας βοηθούν και μας βοηθούν και πριν τις εκλογές στο να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει από χώρα σε χώρα και τι όψη θα έχει το Κοινοβούλιο σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Γιατί, γιατί ε, είναι χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες το βράδυ των εκλογών για να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα και να είμαστε σε θέση να δώσουμε στους πολίτες κάτι το ακριβές πριν ε, λάβουμε τα τελικά αποτελέσματα. Δηλαδή αν ε, περιμένουμε τα 100% των αποτελεσμάτων σημαίνει πως θα περιμένουμε μέχρι Δευτέρα ή και την Τρίτη γιατί κάποιες χώρες είναι κάπως αργές στην ε, καταμέτρηση και την δημοσίευση. Οπότε πρέπει να έχουμε κάποια μερικά αποτελέσματα τα οποία θα μπορέσουμε να μεταφράσουμε σε κάτι πολιτικά κατανοητό για τους μουσιογράφους το βράδυ των εκλογών, ίσως κάπως αργά λόγω του ότι οι κάλπες ε, στην Ιταλία κλείνουν 11 το βράδυ, αλλά τουλάχιστον ε, την ημέρα των εκλογών. Εάν δείτε την προβολή αυτή και εάν δείτε και στο site μας ε, τις προηγούμενες προβολές θα δείτε πως υπάρχουν κάποιες τάσεις που είναι σταθερές εδώ και κάποιους μήνες. Θα περιγράψω λοιπόν κάποιες τάσεις και μια πολιτική ερμηνεία, αν θέλετε, των τάσεων αυτών. Πρώτα απ' όλα βλέπετε πως υπάρχουν δύο πολιτικές ομάδες που είναι λίγο πολύ ε, ισοδύναμες. Τσίμα-τσίμα ε, θα λέγαμε. Δεν θα ξέρουμε μέχρι τις εκλογές βεβαίως, αν ήταν σήμερα θα λέγαμε πως ε, έχουν λίγους ε, παραπάνω βουλευτές έχει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα από τους Σοσιαλιστές αλλά βεβαίως η προβολή αυτή έγινε με δεδομένα που μας ήρθαν πριν ε, ξεκινήσει ουσιαστικά η προεκλογική εκστρατεία. Οπότε ας δούμε το τι θα συμβεί με τις ε, προβολές που θα δημοσιεύσουμε ε, αύριο βράδυ, πέμπτη πρωί το αργότερο. Βλέπετε πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα. Εάν το συγκρίνεται με το τωρινό κοινοβούλιο σημαίνει πως χάνει αρκετούς βουλευτές για τώρα είναι γύρω στους 285 και στην περίπτωση αυτή θα ήταν 215 10 παραπάνω από τους σοσιαλδημοκράτες κάτι το οποίο σημαίνει περισσότερους βουλευτές αλλά τουλάχιστον μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στη δεύτερη θέση οι σοσιαλδημοκράτες. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά ενδιαφέρον είναι ε, να συγκρίνουμε και με το τωρινό κοινοβούλιο. Αν προσθέσουμε τις δύο αυτές ομάδες, ε, το μέγεθός τους θα έλεγα μειώνεται. Τώρα είναι γύρω στο 65%. Οπότε όταν συμφωνήσουν αυτές οι δύο ομάδες σημαίνει πως 65% των βουλευτών στην Ολομέλεια κατά κανόνα θα την υπερψηφίσουν. Στην περίπτωση αυτή το άθροισμά τους μειώνεται από το 65% στο 55% χοντρικά. Σημαίνει βεβαίως απόλυτη πλειοψηφία, αλλά Σημαίνει πως ε, και για να είμαστε σίγουροι πως θα περάσει μια σημαντική ψηφοφορία στην Ολομέλεια πρέπει να είμαστε σίγουροι πως οπωσδήποτε όλοι οι βουλευτές θα είναι στην αίθουσα και βεβαίω πως υπάρχει και εσωτερική πειθαρχία. Αν ξεκινήσουμε να χάνουμε ανθρώπους λόγω της θέσης μιας εθνικής αντιπροσωπείας ή λείπει κάποιος και χρειάζονται 376 για να περάσει κάτι, ε, πρέπει να είμαστε σίγουροι πως ε, το 55% δεν θα γίνει 49% ή 45% την ώρα της ε, ψηφοφορίας. Οπότε τέλος πάντων προβολή είναι αυτό, θα δούμε τι θα γίνει στις 25 του μηνός, αλλά είναι ενδιαφέρον στοιχείο γιατί θα παίξει και ένα ρόλο στις αποφάσεις για το ποιος θα είναι ο επίσημος υποψήφιος για πρόεδρος της Κομισιόν μετά το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να παρακολουθήσουμε προσεκτικά, όχι μόνο σήμερα αλλά και στις 25, είναι πόσους πιθανούς ε, συνδυασμούς συμμαχίες δηλαδή έχουμε με αυτά αποτελέσματα. Υπάρχει, αν θέλετε, η πιθανότητα του μεγάλου συνασπισμού, αν δείτε το τι γίνεται και στο Βερολίνο, ε, μπορούμε να προσθέσουμε βεβαίως και άλλες πολιτικές ομάδες, ε, φιλελεύθερους, πράσινους, αναλόγως του αν ε, σκέφτεται κανείς να εκλέξει πρόεδρο της Κομισιόν ή να περάσει κάποιο νομοθέτημα. Ε, εάν μιλάμε για την οικονομία μπορεί το ΕΛΚ να σκεφτεί τη συνεργασία με τους φιλελεύθερους ή αν μιλάμε για το κοινωνικό μοντέλο οι φιλελεύθεροι να συνεργαστούν με τους σοσιαλδημοκράτες ή τους πράσινους. Έτσι συμβαίνει τώρα τουλάχιστον. Τώρα υπάρχουν λοιπόν τρεις πιθανές ε, συμμαχίες που λειτουργούν και λειτουργούν στην Ολομέλεια. Οι πρώτη είναι σοσιαλιστές, είναι Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ή το κάθε ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα μόνο του ή μαζί με άλλο κόμμα. Το, η άλλη πιθανότητα είναι κέντρο αριστερός, δηλαδή σοσιαλδημοκράτες, φιλελεύθεροι και πράσινοι και καμιά φορά κάποιοι βουλευτές ε, από την αριστερά της αριστεράς, ε, την ε, Ενωμένη Ευρωπαϊκή Αριστερά όπως λέγεται, την ΚΟΕ. Π.χ. αυτός ο συνασπισμός απέρριψε τη συνθήκη για τα δεδομένα SWIFT με τις Ηνωμένε Πολιτείες ή νομοθεσία που αφορούσε στην ιδιωτική ζωή, προστασία προσωπικών δεδομένων κτλ. Αλλά υπάρχει και ένας τρίτος πιθανός συνασπισμός, ο κεντροδεξιός, δηλαδή Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, συμφιλελεύθερη, συντηρητική η ε, Ευρωπαϊκή Συντηρητική δηλαδή κατά βάση είναι η Άγγλη Συντηρητική και κάποιοι Πολωνοί, το κόμμα του Κατσίνσκι στην Πολωνία ε, υπήρχε μέχρι τώρα η δυνατότητα να δημιουργηθεί μια τέτοια πλειοψηφία που δημιουργήθηκε π.χ. για ε, νομοθεσία που αφορούσε τα οικονομικά. Όχι πάντα, αλλά μερικές φορές. Με την προβολή αυτή, αν κάνετε τους υπολογισμούς σας, θα δείτε πόσο μεγάλος ξεκάθα, ε, μεγάλη ξεκάθαρη συμμαχία θα ε, περιέχει τουλάχιστον ε, σοσιαλιστές και ΕΛΚ. Όλοι οι υπόλοιποι δεν φτάνουν το άθροισμα των 376. Και πάλι σας λέω, αυτά είναι προβολές σημερινές με βάση τα όσα δηλώνουν οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες δύο-τρεις εβδομάδες μετά άλλα στοιχεία. Οι μόνες πολιτικές ομάδες ε, είναι, που αυξάνουν τη δύναμή τους είναι στα αριστερά. Σοσιαλδημοκράτες ε, και γκούε. Η αριστερά της αριστεράς θα λέγαμε. Που ε, αυξάνουν ναι. ποσοστιαία περισσότερο τη δύναμή τους από τις άλλες ομάδες. Και αν δείτε τις υπόλοιπες ομάδες ε, μειώνονται ή παραμένουν σταθερές. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, συντηρητική και ίσως η Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας ε, με επικεφαλή στον Νάιτζελ Φάραντζ, το UKIP, ε, τον πρόεδρο του UKIP. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα δύο ενδιαφέροντα στοιχεία, το τι θα συμβεί με τους ε, μη ε, εγγεγραμμένους ε, και τους λοιπούς. Οι μη εγγεγραμμένοι είναι από κόμματα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα μέλη τους δεν ανήκουν σε κάποια πολιτική ομάδα όπως παραδείγματο χάρη το Εθνικό Μέτωπο της Γαλλίας έχει τρεις βουλευτές αυτή τη στιγμή δεν ανήκουν σε κάποια πολιτική ομάδα είναι μη εγγεγραμμένοι όπως λέμε κάτι το οποίο σημαίνει στο 5% αυτό έχουμε μεταξύ άλλων τους βουλευτές που αναμένουμε από το Front National το Εθνικό Μέτωπο της Γαλλίας το ίδιο και στην Ισπανία με το UPD. Ένα κόμμα το οποίο έχει έναν ευρωβουλευτή αυτή τη στιγμή, πάλι είναι στους μη εγγεγραμμένους, οπότε οι βουλευτές που αναμένουμε από το Ιόν Προγκρέσο είναι η Δημοκρασία αυτή τη στιγμή πηγαίνουν στους μη εγγεγραμμένους που θα είναι λίγο πολύ 5% των ευρωβουλευτών και μετά βλέπουμε δύο γκρίζες ζώνες στα δύο άκρα που είναι λυπή. 68 ε, ευρωβουλευτές από πολιτικά κόμματα που ε, δεν ε, προσωπούνται αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράδειγμα προφανές ε, το κίνημα των πέντε αστέρων, το κόμμα υπό την ηγεσία του Μπέπε Γκρίλο. Δεν εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο, δεν ε, ξέρουμε για αν θα ενταχθούν σε κάποια πολιτική ομάδα. Ίσως, ίσως όχι. Αναλόγως λοιπόν. μπορεί να πάνε σε άλλη ομάδα μπορεί να μην ενταχθούν. Μην ξεχνάτε πως για να ε, μπει κάποια ομάδα βεβαίως πρέπει να θέλει αλλά πρέπει και να τον θέλει η ομάδα αυτή. Δεν μπορεί κάποιος να αποφασίσει μόνος του ότι ανήκει σε αυτή την πολιτική ομάδα να πάει στο, στο ΕΛΚ και ας πούμε στους Ευρωπαϊκούς Συντηρητικούς αν δεν τον θέλουν πρέπει και να σε δεχτεί και αυτή η πολιτική ομάδα και σε κάποιες ε, περιπτώσεις ε, αυτό είναι ας πούμε μια απόφαση η οποία δεν λαμβάνεται εντελώ ελεύθερα αλλά ακολουθείται το καταστατικό της κάθε πολιτικής ομάδας. Έχουμε λοιπόν τους λοιπούς σε δύο κομμάτια όπως είπα δεν σημαίνει οπωσδήποτε αριστερά ή δεξιά κάποιοι θεωρούνται ε, αριστεροί άλλοι θεωρούνται δεξιοί οπότε το κόψαμε στην μέση ας πούμε και το 9% αυτό δεν σημαίνει 9% ε, με τον ίδιο στόχο ή με την ίδια ιδεολογία και άρα δεν σημαίνει ότι είναι ένα συμπαγές 9%. Και τελευταία πληροφορία, κάτι το οποίο γνωρίζετε πια, για να δημιουργηθεί νέα πολιτική ομάδα και να διατηρηθεί οπωσδήποτε χρειάζονται τουλάχιστον 25 ευρωβουλευτές από τουλάχιστον 7 χώρες. Ένα τέταρτο των χωρών, δηλαδή 7 αυτή τη στιγμή και αυτό είναι επίσης ενδιαφέρον και θα το δούμε την βραδιά των εκλογών. Πρώτα απ' όλα το τι θα συμβεί με τις ομάδες ε, που ήταν μικρές στο κοινοβούλιο. Αυτό στη τι αυτή, όπως η ομάδα ε, της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας του κυρίου Φάρατς, δεν ξέρουμε αν θα έχει 25 βουλευτές από 7 χώρες. Είναι μια πρόκληση αυτό, οπωσδήποτε, και τι σχέση έχει μετά αυτό με την ύπαρξη ή μη μιας νέας πολιτικής ομάδας ε, που μπορεί να δημιουργηθεί από την ε, άκρα δεξιά. Και ξέρετε επειδή παρακολουθούμε την ομάδα αυτό θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της Μαρίν Λεπέν ή του κυρίου Βίλντερς ε, στην Ολλανδία και άλλων σε άλλες χώρες αλλά και πρέπει να δούμε βεβαίως το αν έχουν 25 βουλευτές που θα είναι εύκολο κατά την άποψή μου αλλά το εάν οι 25 αυτοί βουλευτές ε, ε, προέρχονται από τουλάχιστον 7 κράτη-μέλη και όσον αφορά δε την ε, δυνατότητα, την πιθανότητα μια ομάδας στα ακροτεξιά αυτό θα έχει συνέπειες και για την ομάδα της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας του κυρίου Φάρατζ. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν θα υπάρχουν αρκετοί βουλευτές για 8 ή για 7 ομάδες όπως τώρα. Όπως και στην προηγούμενη θητεία. Θα σταματήσω. Εδώ νομίζω σας έδωσα τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία. Και βεβαίως καλό είναι να παρακολουθείτε τις επόμενες προβολές, ε, η επόμενη μάλλον αύριο το απόγευμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορούμε να συνεχίσουμε με κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις. Δυστυχώς η διερμηνία πρέπει να σταματήσει τώρα, αλλά μπορείτε να εκφραστείτε στα αγγλικά και να ακούσετε αγγλικά. Σταματάει τώρα